Bueno, vamos eh, Ας αρχίσουμε. Αρχίζουμε με το πρώτο τμήμα. Όσον αφορά τις αποστολές δηλαδή στην Τουρκία που πήγε εκεί η επιτροπή μας και την συμμετοχή μας στην παγκόσμια ανθρωπιστική διάσκεψη και μετά θα περάσουμε στην ακρόαση για τις μειονότητες. Ανάμεσα στη Συρία και το Ισλαμικό λεγόμενο κράτος, στο Ιράκ κλπ. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν λίγες στην ημερήσια διάταξη, προχωράμε. Εντάξει αν δεν διαφωνεί κανείς, να εγκρίνουμε και τα πρακτικά της 3ης ε, ε, Μαρτίου και του Απριλίου. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τρία κατεπήγοντα στο Στρασβούργο που μας πέρασε όσον αφορά τους Σταρτάρους στην Κρυμαία, την Κάμπια και το Τζιμπουτί. Επίσης, συζητήθηκαν και άλλα θέματα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την ε, υποπιτροπή μας. Για παράδειγμα, αυτό που έχει να κάνει με την οδηγία για την ε, πρόληψη εμπορίας ανθρώπων και πώς θα προστατευτούν τα θύματα, λαμβάνοντα υπόψη την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όσον αφορά την Τουρκία τώρα συγκεκριμένα, έχουμε εδώ πέρα δύο στοιχεία. Το ένα είναι το ταξίδι, δηλαδή η αποστολή της δικιάς μας υποπιτροπής που πήγε στην Τουρκία 16 με 18 Μαΐου. Στόχος της επίσκεψης αυτής, τη αποστολή αυτή ήταν να εξετάσει την κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και στα πλαίσια τη συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία. Έχουμε μαζί μας την κυρία Σχάκε και τον κύριο Λίτς, που είναι δύο μέλη της υποπιτροπής αυτής που συμμετείχαν σε αυτήν την αποστολή. Γι' αυτό και θα του δώσω το λόγο. Παρακαλώ, κυρία Σχάκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε να μοιραστώ μαζί σας τις εμπειρίες μας από την επίσκεψή μας αυτή, η οποία έγινε σε κάποια πολύ σημαντική στιγμή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίως και είπε τη γνώμη του, ποιες είναι οι ανησυχίες μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου κλπ. κλπ. Και είχαμε πολλούς λόγους να ανησυχούμε τα τελευταία χρόνια για αυτά. Και ήταν ξεκάθαρο κατά τη διάρκεια της ε, επίσκεψής μας εκεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, επιφέρει περισσότερες κριτικές από ό,τι ίσως Κομισιόν και το Συμβούλιο, κυρίως μετά από τη συμφωνία για, την, ε, το μετασταυτικό και το προσφυγικό. Παραβιάσεις κράτους δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερία του τύπου, η κατάσταση των προσφύγων εκεί, και μάλιστα σε σχέση με τους πρόσφυγες, κυρίως για την κατάσταση των γυναικών και των παιδιών προσφύγων, που είναι και η πλειοψηφία των προσφύγων εκεί. Κοιτάξαμε επίσης τι γίνεται και με το ΠΚΚ και τα τουρκικά στρατεύματα, τα οποία δυσανάλογα έχουν χτυπήσει τους αμάχους ε, εκεί. Μισό εκατομμύριο από αυτούς από ό,τι φαίνεται έχουν αναγκαστεί να μετατοπιστούν. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο δεν ακούγεται συχνά εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι όμως πολύ σημαντικό. Κατά την επίσκεψή μας αυτή, δύο ημερών, συζητήσαμε με διεθνείς οργανώσεις εκεί, με κόσμο που δουλεύει μαζί τους τη UNICEF, με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Διατροφής, με τουρκικές οργανώσεις και με κυβερνητικές που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τους πρόσφυγες, αλλά και με διεθνείς μη κυβερνητικέ οργανώσεις που δουλεύουν εκεί στην Τουρκία. Μιλήσαμε και με ακαδημαϊκούς. Μία γυναίκα η οποία χάσε τη δουλειά της επειδή υπέγραψε ένα κείμενο για συλλογή υπογραφών που είχε να κάνει με υπουργούς που είχαν ε, αναγκαστεί να φύγουν. Ε, μιλήσαμε και με ομολόγους μας από το και, και άλλα βασικά κόμματα στην Τουρκία και Μιλήσαμε και με το ΧΑΝΤΕΠΕ και τον επικεφαλής. Τη μέρα ακριβώς που στο τουρκικό κοινοβούλιο συζητούσαν την άρση ασυλίας των βουλευτών στην Τουρκία, στην ε, Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Έγινε μία unblock ψηφοφορία που οδήγησε σε μία κατάσταση όπου 130 βουλευτές, όπου υπάρχουν ε, εναντίον τους ε, κατηγορίες, συγκεκριμένα για το HDP είναι 50 από τους 59 βουλευτές εναντίον των οποίων υπάρχουν κατηγορίες. Ήταν δηλαδή μια πολύ βασική στιγμή, σημαντική στη ζωή του Κοινοβουλίου της ε, Τουρκίας και επίσης ήταν και το θέμα της εκλογής του νέου Πρωθυπουργού. Ένα βασικό ζήτημα που συζητήσαμε ήταν η ελευθερία του τύπου. Αυτή είναι μια μεγάλη ανησυχία εδώ και χρόνια, όπω επίση η ελευθερία στο διαδίκτυο. Συναντηθήκαμε με δημοσιογράφου από τρει εφημερίδε και είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε και με τον Τζον Ντούνταν, ο οποίο είναι δημοσιογράφο, ο οποίο έχει καταδικαστεί σε πέντε χρόνια φυλακή, περιμένει το αποτέλεσμα τη Έφεση και αυτό γιατί δημοσιοποίησε μια υπόθεση που είχε να κάνει με, όπως λένε, κρατικά μυστικά. Και υπήρξε και υπήρξε κατά τη ζωή του την ημέρα που βγήκε η απόφαση. Είναι σημαντικές στιγμές αυτές στη ζωή της Τουρκίας. Τέλος, που καταλήξαμε. Εμείς εδώ πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τα εξή. Α, να προσθέσω και ότι συναντηθήκαμε και με τον διαμεσολαβητή, τον συνήγορο του πολίτη δηλαδή εκεί στην Τουρκία μερικές φορές στα χαρτιά υπάρχουν οι νόμοι. Δηλαδή υπάρχει ο θεσμός του συνήγορου του πολίτη. Συχνά όμως το γράμμα του νόμου δεν είναι το ίδιο με αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα. Βλέπουμε δηλαδή να εφαρμόζεται αυθαίρετα ο νόμος πολλές φορές, να επηρεάζεται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται ο νόμος, να μην υπάρχει όπως θα έπρεπε διάκριση εξουσιών και ακόμα και οι θεσμοί μερικές φορές δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Αυτό πρέπει να προσέξουμε πιο πολύ. Δηλαδή, έχει μόνο τι υπάρχει στο χαρτί, υπάρχουν οι θεσμοί, υπάρχουν οι ρήτρε ασφάλεια κτλ. Αλλά στην πράξη να δούμε τι γίνεται. Είναι επίση σαφέ ότι η ελευθερία του τύπου και η πόλωση στην κοινωνία έχει οδηγήσει σε μεγάλες εντάσεις μεταξύ των θεσμών, μεταξύ των ανθρώπων του κόσμου και των θεσμών και θα έλεγα ότι υπάρχει και ένα κλίμα φόβου μεταξύ πολλών ανθρώπων στη χώρα. Σε μια κατηγορία δηλαδή του πληθυσμού. Τώρα όσον αφορά αλλαγέ για την νομοθεσία κατά της τρομοκρατίας από βλέπεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι αλλαγές αυτές θα είναι πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές στην ευρωπαϊκή αυτή νομοθεσία στην Τουρκία αποτελούν μέρος των απαιτήσεων τα όσα συμφώνησαν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία και οι δύο το 2013 για μεταρρυθμίσεις δηλαδή οι οποίες πρέπει να γίνουν ώστε να επιτραπεί η κατάργηση της θεώρησης της βίζα για τους Τούρκους πολίτες. Τώρα λοιπόν βιαζόμαστε εξαιτία της συμφωνίας αυτής για το μεταναστευτικό για το οποίο η Τουρκία ζητάει αυτή την κατάργηση της θόρησης. Πρέπει να δούμε όμως ακόμα τι αλλαγές θα γίνουν στον αντιτρομοκρατικό νόμο. Πολλά διακυδεύονται εδώ και πολλοί θα πούνε ότι ο νόμος, μάλλον ότι η συμφωνία πρέπει να περάσει όπως και να έχουν τα πράγματα. Πάντως εμείς αυτό που διαπιστώσαμε εκεί είναι ότι η νομοθεσία κατά της τρομοκρατίας χρησιμοποιείται για να σωπαίνουν οι φωνές επικρίσεων εξαιτία θεμάτων ε, εθνική ασφάλειας και τα λοιπά. Σαν άλλο θα χρησιμοποιείται η νομοθεσία αυτή. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται μόνο για τις παραβιάσεις στο νοτιοτολικό τμήμα της Τουρκίας που πρέπει να μας απασχολεί όλους δεδομένων νέων ροών προσφυγικών αλλά και των εντάσεων που έχουμε στα σύνορα στη Μέση Ανατολή αλλά και επειδή ο αντιτρομοκρατικός νόμος χρησιμοποιείται για να σωπούν οι επικρίσεις, να μην ακούγονται. Θα έπρεπε να γίνεται η συζήτηση, η δημόσια συζήτηση πιο ζωντανά, πιο ελεύθερα. Και οι πολιτικές αλλαγές να στηρίζονται από τον κόσμο. Αυτά προς το παρόν. Τώρα, αν οι συνάδελφοι θέλουν κάποιες λεπτομέρειες, ευχαρίστως. Έπειτα είναι εδώ και οι συνάδελφοι. Σίγουρα ήταν μια συνάντηση με πολλά δυνατά, πολλές δυνατές στιγμές. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριος Λίτς. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θέλω καταρχάς να ευχαριστώ την κυρία Σχάκια για την ε, οργάνωση και την εποπτεία στη λειτουργία της ομάδας μας. Τρεις είμαστε, αλλά μπορέσαμε να οργανωθούμε τους να καλύψουμε πολύ υλικό και ευχαριστώ και τη γραμματεία. Ήταν πολύ εντατική η επίσκεψη. Είχαμε 9-10 συνεδριάσεις μέσα σε μία ημέρα και καθοδόν ακόμη. Και από αυτά που υπόθηκαν δεν θέλω να επαναλάβω τίποτα. Θέλω θα, μόνο να σημειώσω όταν είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εξέλιξη Εκείνη τη εβδομάδα και σε σχέση με τα θέματα των μέσων ενημέρωση, ε, την απελευθέρωση τη ε, υποχρέωση θεώρηση διαβατηρίου. Πολλέ φορέ ε, ρωτηθήκαμε για τα θέματα αυτά. πολλοί και πανεπιστημιακοί αλλά και κοινοί πολίτες χίλιοι τουλάχιστον ήταν αυτοί οποίοι έχουν υπογράψει μια δήλωση όπου ζητούν κατάπαυση πυρός στην Ανατολική Τουρκία και απελήθησαν στη συνέχεια από τις θέσεις τους, ακόμα και πανεπιστημιακοί. Εγώ θα έλεγα ότι προχωρούμε πλέον προς μια δικτατορική μορφή διακυβέρνησης, προεδρική δικτατορία θα την ονόμαζα, εάν δεν προσέξουμε, γιατί οι εξελίξεις είναι ταχύτατες. Και από τα κοινοβουλευτικά ε, κόμματα με τα οποία συναντηθήκαμε το ΧΑΝΤΑΠΕ δείχνει μεγάλη ανησυχία από τους 59 ή 50 βουλευτές του ε, έχουν ε, την απειλή της ποινικής δίκησης βάρος τους και οι δίκες που έχουν γίνει με μήνυση του ίδιου του Προέδρου είναι ασύγκριτα σε σχέση με χώρες πολλές. Πρέπει λοιπόν να εκδηλώσουμε αμέριστη συμπαράσταση πλέον. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες δικών σε εξέλιξη, όχι μόνο εις βάρος πανεπιστημιακών δασκάλων, αλλά και άλλων δημοσιογράφων, εργαζομένων στο μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικότερα, όπως είπαμε. Και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην Τουρκία πλέον. Και λόγω της σημασίας που έχει από κοινού να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή. Πολύ συχνά λέγεται ότι έχει κάνει πολλά για να βοηθήσει στην περίπτωση των προσφύγων η Τουρκία. Είχαμε γενική αποτίμηση από τη συνάντησή μας με τη UNICEF και την Υπατή Αρμοστία και μας είπαν ότι είναι το χαμηλότερο επίπεδο ε, αυτό που βλέπουν στην Τουρκία σε σχέση με παρουσία ε, μη, κυβερνητικών οργανώσεων, ενώ στις ε, αφρικανικές χώρες έχουν μεγάλο πεδίο δράσης. Στην Τουρκία είναι πολύ περιορισμένη η δράση τους. Στην Τουρκία 46% των προσφύγων είναι παιδιά και πέραν αυτών οι περισσότεροι γυναίκες πρόσφυγες. Και έτσι η διάθεση κονδυλίων θα πρέπει να στρέφεται όχι προς την τουρκική κυβέρνηση, αλλά προς τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις να στηρίξουμε το έργο τους, εάν πρόκειται να διατεθούν περισσότερα κονδύλια από την ευρωπαϊκή πλευρά. Αφού συναντήσαμε τον κύριο Τζουντάρ, που μας είπε ότι θα ήταν σκόπιμο να γίνουν ε, άλλες συναντήσεις με υποστηρικτές. Θα πήγαινε μάλιστα και η Μέρκελ ε, στην ε, Τουρκία και εν ώψη αυτής της επίσκεψης της ε, κρίθηκε σκόπιμο να πιέσουμε εμεί από πλευρά μα για να συναντήσει τον Τζουντάρ η Μέρκελ, πράγμα το οποίο δεν υλοποιήθηκε τελικά. Από εφημεριδε η ίδια η Χουριέτ απειλείται. Ε, αν και ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί αυτή η απειλή, πάντω υπάρχει, είναι ορατή. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφεί, απερίφραστοι ω κοινοβούλιο και να μην κάνουμε την παραμικρή υποχώρηση σε σχέση με τις 72 προϋποθέσεις για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης. Είτε ο πρόεδρος στη Γερμανία, όποιος είναι να λάβει αποφάσεις, δεν πρέπει να αφήσει κανένα περιθώριο και να κάνει οδήποτε συμβασμό σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πέραν αυτών, θέλω να υπογραμμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισκέπτεται την Τουρκία τον Ιούλιο. Δεν ξέρω εάν η Επιτροπή μας εμπλέκεται σε αυτόν, θα πάει κάποιος δικός μας συνάδελφος αλλά πάντως πρέπει να φροντίσουμε οι συνάδελφοι που θα επισκεφθούν με την αντιπροσωπή αυτήν ε, να ακούσουν τις δικές μας θέσεις και να τους παρακαλέσουμε να μας μεταφέρουν ό,τι οι ειδήσει αποκομίσουν από εκεί, γιατί σκοπεύουν να πάνε και στην νοτιοανατολική χώρα, από ό,τι φαίνεται, όπου έχουμε να κάνουμε με εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες οι οποίοι είναι διάχυτοι στην Τουρκία και δεν ε, την χάνουν της υποδοχής ε, που θα χρειάζονταν. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς. Κι εγώ ήθελα να προσθέσω κάτι στα όσα είπαν οι δύο συνάδελφοι. Παρόλο που θα τα δούμε βέβαια και στη συνέχεια όταν θα αναφερθούμε στην ανθρωπιστική διάσκεψη. Στην επίσκεψή μας στην Κωνσταντινούπολη πάντως, για την διάσκεψη αυτή. Είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με πολύ κόσμο, είτε από τα μέσα ενημέρωση, είτε από οργανώσεις, μη κυβερνητικέ οργανώσεις γυναικών κλπ. Και έτσι, εγώ διαπίστωσα ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία, όπως ακριβώς είπαν και οι συνάδελφοι. Υπάρχει δηλαδή μία σαφής καταπίεση. Έχουμε πολλά στοιχεία που μας γίνουν ανησυχίες. Η κατάσταση στην Τουρκία είναι δύσκολη. Έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί. Αλλά αυτό δεν φτάνει για να τα εξηγήσει όλα. Η εντύπωσή μου δηλαδή είναι ότι η θέση μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι δύσκολη. Γιατί από τη μια δεν πρόκειται βέβαια να εγκαταλείψουμε τον τουρκικό λαό, ο οποίος είναι σαφές ότι θέλει να έρθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη μεριά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για την κατάσταση, δηλαδή για την έλλειψη ελευθεριών και γενικά για όλα τα βήματα που κάνει προς τα πίσω η Τουρκία, όσον αφορά τις γυναίκες για παράδειγμα αλλά όχι μόνο. Η νομοθεσία ίσως να μην περάσει πριν το καλοκαίρι, αλλά προβλέπεται μια νομοθετική τροποποίηση η οποία κάνει διαφορά ανάμεσα στις γυναίκες τις παντρεμένες και τις ανήπεντρες σε σχέση με τα κοινωνικά επιδόματα κτλ. Υπάρχει θέληση της κυβέρνησης να υποστηρίξει τις οικογένειες, εντάξει, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια διάκριση. Όπως είπανε και οι συνάδελφοι, μιλήσαμε επίσης και με πολλούς σημαντικούς δημοσιογράφους. Έχουν κλείσει εφημερίδες, διώκονται ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι. Αυτό είναι κάτι συνηθισμένο, καθημερινό φαινόμενο εκεί. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι πιστεύω πως το Κοινοβούλιο πρέπει να παραμείνει σε γρήγορση και να παρακολουθεί την διαδικασία εκεί, η οποία από δημοκρατική άποψη μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Δεν έχει να κάνει με το αν αναγνωρίζουμε την αλληλεγγύη της Τουρκίας ή όχι απέναντι στους πρόσφυγες. Μπορεί κανείς να είναι αλληλέγγυος προς τους πρόσφυγες, αλλά να καταπιέζει το λαό του. Έτσι, γίνεται αυτό. Συνεπώς, αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι ενισχύουμε ιδιαίτερα για τα αρνητικά τα οποία εντοπίσαμε και διαπιστώσαμε στις διάφορες μετακινήσεις μας ανά τη χώρα. Μία αντιπροσωπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επίσημη, κατά πάσα πιθανότητα τον Ιούλιο θα πάει εκεί, υπό την μόνιμη συγγητριά μας, την Κάτι Πύρη, που γνωρίζει βέβαια πάρα πολύ καλά τόσο τη χώρα, όσο και τις ανησυχίες μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και μαζί της τότε. Τώρα, εκπρόσωπος της πρεσβείας της Τουρκίας έχει ζητήσει το λόγο Αϊσέισερ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. και τη δυνατότητα που μας δίνεται να σχολιάσουμε αυτή την επίσκεψη. Από ό,τι γνωρίζουμε αυτή η επίσκεψη κάλυψε μια, ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και προσέφερε καλή ευκαιρία για συναντήσεις με αρχές τουρκικές εκπροσώπους των, της κοινωνίας των πολιτών. Από ό,τι γνωρίζω είχατε επικοινωνία με διάφορους εκπροσώπους τομέων, ε, είτε από την κυβέρνηση, με κυβερνητικές οργανώσεις. Και θεωρούμε ότι είναι καλό αυτό, γιατί προσφέρει πολύ χρήσιμες και καρποφόρες ανταλλαγές απόψεων, χρήσιμες συζητήσει που πιστεύουμε είναι ουσιώδους σημασία για τις σχέσεις μας. Μπορεί να ανοίξει έτσι ένας ειλικρινής διάλογος, μια επικοδομητική προσέγγιση ως βάση αυτών των σχέσεων. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ πρώτα στη μετανάστευση. Όλοι γνωρίζουμε βεβαίως ότι η Τουρκία είναι η μόνη χώρα στον κόσμο, αν κοιτάξετε τα νούμερα, των παράτυπων μεταναστών, Είμαστε η χώρα που έχει τον υψηλότερο αριθμό παράτυπων μεταναστών. να πριν πλέον στα 3 εκατομμύρια. Μόνο 10% των μεταναστών, λέει ο Μιλήτρια, ζουν σε καταβλισμούς. Όλοι οι υπόλοιποι είναι διασπαρμένοι ανά τη χώρα. Με την ανάδειξη της μεταναστευτικής κρίσης, έλαβαν νέα δυναμική κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Άνοιξε μια νέα σελίδα, γυρίσαμε σελίδα, μια δυναμική που θέλουμε να διατηρηθεί. Και με βεβαία ότι γνωρίζετε και εσείς πως η συμφωνία της 18ης Μαρτίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας λειτουργεί πολύ καλά. Οι παράτυποι μετανάστες που διασχίζουν τον ε, το Αιγαίο, το Φεβρουάριο ήταν 850. Στο Μάιο ο μέσος όρος έχει πέσει στους 20. Τεράστια επιτυχία λοιπόν. Κανείς δεν μιλάει πλέον για υπαρξιακή κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πια. Και μπορούμε υπερήφανα να πούμε ότι έφεραν καρπούς οι προσπάθειές μας, οι κοινέ μας προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα. Τις υποσχέσεις μας τις στηρίσαμε και τις στηρούμε στο πλαίσιο των συμφωνιών. Έχουμε δεχθεί μέχρι τώρα τα 341 παράτυπους μετανάστες από την Ελλάδα, εκ των οποίων μόνο 18 είναι Σύριοι, υπήκοοι, οι περισσότεροι είναι Πακιστανοί, η Γερμανία, οι κάτω χώρες, η Λιθουανία, η Σουηδία έχουν μέχρι τώρα υποδεχθεί 319 Σύρους Όπως είπα, εμείς τις υποσχέσεις μας τις στηρούμε και αναμένουμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να πράξει το ίδιο βάσει της συμφωνίας μας. Απελευθέρωση δηλαδή της θεωρής διαβατηρίων και οικονομική υποστήριξη για τους Σύρους. Θέλω εδώ να υπογραμμίσω ότι αυτή η οικονομική υποστήριξη δεν πηγαίνει, δεν κατευθύνεται στην ε, τουρκική κυβέρνηση, αλλά το συριακό πληθυσμό στην Τουρκία. Μια άλλη υπόσχεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά το άνοιγμα νέων κεφαλαίων. Για τη θεώρηση διαβατηρίων το μεταξύ θέλω να πω ότι ναι, έχετε δίκιο πως υπάρχουν 72 κριτήρια που πρέπει να εκπληρωθούν, όπως συμβαίνει για κάθε χώρα. Θα, τις θα τα εκπληρώσει η Τουρκία. Ο κύριο Τίμερμαν, πρώτο αντιπρόεδρο, όπω γνωρίζετε, ασφαλώ επισκέφθηκε την Τουρκία την ε, προηγούμενη Παρασκευή για διαπραγματεύσει με Τούρκου αξιωματούχου. Εξ όσων γνωρίζω, έχουν καταλήξει σε συμφωνία, χωρί να γνωρίζω τι λεπτομέρειε τη όμω. Υπάρχει συμφωνία. Το ΔΕ Συμβούλιο της Ευρώπης ε, είναι διατεθειμένο να μας ε, υποστηρίξει σε σχέση με τον αντιτρομοκρατικό νόμο με βάση τους κανονισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την υπόθεση Jean Dundar. Εκκρεμωδική αυτή τη στιγμή. Και σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχει τίποτα άλλο να γίνει παρά να ε, στηριχθούμε στη λειτουργία του δικαστικού συστήματος για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, δεν θέλω να πω επίσης δύο λόγια. Η Τουρκία αγωνίζεται διαρκώς κατά της τρομοκρατικής απειλής, χρόνια τώρα. Είμαστε αποφασισμένοι να εκριζώσουμε την τρομοκρατία και χωρίς να θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Από τον Οκτώβριο του 2015, 550 Τούρκοι αξιωματικοί και δημόσιοι λειτουργοί έχασαν τη ζωή τους στις περιοχές όπου σοβεί η τρομοκρατία. Και θέλω να υπογραμμίσω πως η τουρκική κυβέρνηση αγωνίζεται όχι κατά του κουρδικού πληθυσμού, αλλά κατά της τρομοκρατίας του ΠΚΚ στην Νοτιοανατολική Τουρκία. Ευχαριστώ. Sí, señor Henkel. Henkel, Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σε όσους μετέβησαν στην Τουρκία. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν αναφερθήκατε καθόλου στον ε, αντίκτυπο της ε, Ισλαμοποίησης της ε, Τουρκίας που γίνεται όλο και περισσότερο, κάτι το οποίο έχει ως αντίκτυπο ε, έχει αντίκτυπο και στα δικαιώματα των γυναικών. ποιος είναι ο λόγος δεν το διερευνήσατε, δεν το διαπιστώσατε, ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο δεν ακούσαμε τίποτε σχετικά με αυτό το θέμα στην έκθεσή σας ε, για την επίσκεψη αυτή. Ακούσατε επίσης ε, τίποτε σε σχέση με την παρενόχληση χριστιανών στην Τουρκία. Και το τρίτο ερώτημα που θα ήθελα να θέσω είναι κάτι το οποίο αναφέρθηκε στα μέσα ενημέρωσης ε, ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή αφήνουν μόνο τους πρόσφυγες με χαμηλή, χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης να περάσουν στην Ευρώπη και αυτό για οποιονδήποτε δικό τους ε, λόγο υπόθηκε από την εκπρόσωπο της τουρκικής ε, πρεσβείας ε, ότι ο αριθμός των προσφύγων που περνούν στην Ευρώπη είναι πλέον 20 και είπατε ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Όμως υπάρχει και άλλη στατιστική που λέει ότι ε, μόνο 7 άτομα πνίγηκαν από τότε που άρχισε να ισχύει η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία. Πράγματι, είναι λιγότερο από ό,τι πριν. Αλλά το ερώτημά μου είναι το εξή. Ε, σκεφτήκατε ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι πνίγονταν πιο πριν Θα ήθελα να ε, σας ρωτήσω το εξής. Η διάκριση μεταξύ του τουρκικού λαού και του ΑΚΠ είναι αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε. Έχω πάει πολλές φορές στην Τουρκία, γνωρίζω καλά αυτή την Τουρκία, όπως φαντάζομαι και πολλοί άλλοι. Ε, μπορεί να τη συμπαθείτε, να μην τη συμπαθείτε, αλλά... Ε, είναι πράγματι Ιδιαιτέρως καταθλιπτική η εικόνα και νομίζω ότι στην επικοινωνία μας με την Τουρκία ε, θα έπρεπε όλο και περισσότερο να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ ΑΚΠ και ε, ε, Τούρκων και αυτοί οι οποίοι περισσότερο υποφέρουν λόγω του Ερντογάν δεν είμαστε εμείς αλλά οι ίδιοι Τούρκοι. Ευχαριστώ. Η κυρία Σχάκη και μετά ο κύριος Λίτς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για ε, την ερώτηση, όπως επίσης και για ε, τα σχόλια της ε, εκπροσώπου της τουρκικής πρεσβείας. Είναι προφανές ότι το να μπορέσω να σας δώσω όλε τις λεπτομέρειες μια επίσκεψη διήμερη, σε ε, δύο λεπτά δεν γίνεται. Αυτό είναι ένας περιορισμός που έχουμε και σε δύο μέρες μπορεί να μην μπορούσα να σας τα πω. Κάτι ακόμη για κάποια συγκεκριμένα θέματα που θίξατε. Το πρώτο το γεγονός ότι πραγματικά ε, καταλαβαίνουμε και εκτιμούμε το ρόλο της Τουρκίας όσον αφορά την αντιμετώπιση των, ε, της κρίσης των προσφύγων. Ε, ε, υπήρχε και μάλιστα και μια συμφωνία αποσύνδεσης όλων των υπολείπων θεμάτων που αφορούν την Τουρκία με την, από την ένταξή της και από τα θέματα των προσφύγων. Τώρα το ερώτημα που θέσατε σχετικά με την Ισλαμοποίηση της ε, Τουρκίας, κύριε Χένκελ, δεν είναι ένα θέμα το οποίο ανέκυψε στις συζητήσεις μας με τους συνομιλητές μας. Ε, αυτό το οποίο δημιουργεί μεγάλη ανησυχία στους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλήσαμε και αυτές είναι και οι δικές μου, η δική μου εντύπωση κατά τα τελευταία 15 χρόνια, είναι ότι υπάρχει όλο και περισσότερο ιδιαίτερο η τάση συγκέντρωση τη εξουσία και ελέγχου από πάνω προς τα κάτω, συγκέντρωση τη εξουσίας σε μικρή, σε, σε, σε, σε λίγα χέρια. Ε, υπάρχουν προβλήματα ε, κράτους δικαίου, υπάρχουν ε, προβλήματα ε, εφαρμογής τη νομοθεσίες Υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα και δημιουργούν σοβαρές ανησυχίε. Αυτό ο έλεγχος λοιπόν από, τα, από πάνω προ τα κάτω... Ε, δεν ε, έχει να κάνει κατά πολλού μόνο με το θρησκευτικό κομμάτι. Θεωρούν ότι είναι ένα παιχνίδι εξουσία. Άλλοι έχουν διαφορετική άποψη και τα δύο θα ήταν ανησυχητικά. Αλλά πιστεύω ότι το γεγονό ότι όλο και περισσότερο αυταρχισμό ε, υπάρχει ε, είναι κάτι το οποίο προέκυψε σε όλε τι συζητήσει που κάναμε. Μιλήσαμε για τον αντίκτυπο στι μειονότητε που θεωρήσαμε ότι ήταν ευρύτερο θέμα. Δεν αφορούσε μόνο θρησκευτικέ και εθνοτικέ μειονότητε, αλλά ανθρώπου ε, με διαφορετικές απόψεις. Ε, είναι κάτι το οποίο βρίσκεται υπό απειλή στην Τουρκία και δεν ακούσαμε ε, συγκεκριμένους φόβους να εκφράζονται για παρενόχληση κατά των χριστιανών, όπως αναφέρατε. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Προφανώς ε, μας ανησυχεί η τρομοκρατία. Δεν, φυσικά μας απασχολεί αυτό το θέμα, δεν θα έπρεπε να ε, παραγνωρίζεται, αλλά ούτε θα έπρεπε να γίνεται κατάχρηση αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας. Ακούσαμε επίσης ε, κάποιες αναφορές ότι υπήρχαν κάποιες, ε, γινόταν μια διαλογή των ε, προσφύγων ανάλογα με το επίπεδο της εκπαίδευσής τους, αλλά δεν ακούσαμε τόσες πολλές αναφορές ώστε να χρήζουν κατά τη γνώμη μας περισσότερης έρευνας. Η συμφωνία που έγινε κατά τη γνώμη μου για τους ανθρώπους που φεύγουν από έναν φρικτό πόλεμο θα έπρεπε να παρακολουθείτε και θα έπρεπε και εμείς να διαδραματίζουμε το ρόλο μας. Είναι γεγονός ότι φαίνεται να είναι απλώς μια πολιτική χειραψία. Από τη μία υπάρχουν τεράστιες προσδοκίες και από τις δύο πλευρές για το ε, τι ακριβώς ε, θα καταφέρει η άλλη πλευρά και βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες κατηγορίες και επικρίσεις ε, κάθε μέρα στις εφημερίδες δεν υπάρχει όμως τίποτε γραμμένο, είναι πάρα πολύ αόριστη αυτή η συμφωνία, δεν υπάρχουν σοβαρέ, συγκεκριμένες δεσμεύσεις και αυτό είναι ο λόγος που υπάρχει αυτό. Όλα αυτά τα στοιχεία της σχέσης μας ε, έχουν κατά κάποιο τρόπο ε, παγιωθεί σε αυτή τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας και δημιουργείται η εντύπωση ότι αν κάτι δεν πάει καλά υπάρχει περίπτωση ολόκληρη η σχέση να καταρρεύσει. Αυτό νομίζω ότι είναι αρκετά κοινικό γιατί βλέπω ότι γίνονται κοινικά σχόλια εκατέρωθεν ε, και το γεγονός ότι ε, οι πρόσφυγες έχουν γίνει απλώς διαπραγματευτικά πιόνια είναι πραγματικά ε, ντροπή για ε, την Ευρώπη του 21ου αιώνα. Υπήρχαν επίσης ανησυχίες για τον αντίκτυπο της δημογραφικής εξέλιξης κάποιων περιοχών όπου μία μειονότητα μπορεί να ζει και πολύ πρόσφυγες διαφορετικού, ε, διαφορετικής προέλευσης ε, έχουν τοποθετηθεί εκεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο ίσως θα μπορούσε να διερευνηθεί περισσότερο. Ε, το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχει μια δημογραφική πολιτική σε σχέση με την κατανομή των προσφύγων στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να το προσέξουμε γιατί υπάρχει μια ευάλωτη κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και πρέπει να το προσέξουμε. Όσον αφορά τώρα τη διάκριση μεταξύ της πολιτικής, ε, της κυβέρνησης και, ε, και του πληθυσμού, ε, Προφανώς εμείς δεν μπορούμε να δούμε μια κυβέρνηση ε, μόνη της, προφανώς εκπροσωπεί ε, τους πολίτες. Ε, μπορούμε να κάνουμε βέβαια ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε ότι οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας δεν είναι μόνο μια κατηγορία διακυβερνητικών συμφωνιών. Σίγουρα ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό, σίγουρα μπορούμε το κάνουμε αυτό. Και κύριε Έγκελ, είμαι βέβαιο ότι έχετε μέσα στην καρδιά σας τη χώρα αυτή και αυτό είναι ο λόγο των σχολείων που κάνατε. Νομίζω πάντως ότι μπορούμε να εξακολουθήσουμε να είμαστε ε, ε, ε, δίωδοι επικοινωνίας και ας ελπίσουμε ότι το αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας είναι ότι, θα είναι ότι ε, οι άνθρωποι στην Τουρκία ε, που θέλουν να έχουν μια ευρωπαϊκή προοπτική να μην απογοητευθούν. Θέλουμε να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με την Τουρκία και ενδεχομένως να δούμε και όλας και την ένταξη της Τουρκίας κάποια στιγμή ε, στο άμεσο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην απογοητευθούν οι άνθρωποι που το περιμένουν αυτό να μην ε, χάσουμε την εμπιστοσύνη μας ε, για τη σχέση αυτή που θα μπορούσε να βασίζεται σε συγκεκριμένε αρχέ παρά το γεγονό ότι ε, πολιτικά μπορεί να διαφωνούμε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία συζητήθηκαν κατά τι συναντήσει μα. Είναι αδύνατο να σα πω τα πάντα. Θα μπορούσα για ώρε να μιλώ, αλλά δεν θα το κάνω. Θα ήθελα απλώ να πω ότι αν σα ενδιαφέρει, συνάδελφοι, πριν από την επόμενή μα επίσκεψη, κατά τη διάρκεια τη ε, προετοιμασία τη ψηφοφορία για ε, την απαλλαγή από θεωρήσει, ευχαρίστω να έρθετε μαζί, να, έρθετε να συζητήσετε μαζί μα, να έρθετε σε επαφή μαζί μα. Πάντω είναι μια κρίσιμη χρονική στιγμή και ελπίζω ότι μπορούμε να διαδραματίσουμε το ρόλο μας και να συνεχίσουμε να εστιάζουμε στις ε, αρχές, τις σημαντικές που θα έπρεπε να ε, υποστηρίζουν ε, κατά τη γνώμη μας τη σχέση, τη σχέση μας. Ο κύριος Λίτς. Ευχαριστώ πολύ γιατί, για τα όσα να ακούσαμε και σας ευχαριστώ που μας προσφέρατε και εσείς την δικιά σας οπτική γωνία. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε από την αρχή, στο πού βρισκόμαστε, τι υποστηρίζουμε και για να επανέλθω, γιατί αυτό το πολύ βασικό αυτό που όλοι οι ομολογοί μας μας ε, ζήτησαν και αυτό είναι να επιμείνουμε και να μην απομακρυνθούμε καθόλου από τις επικρίσεις μας όσον αφορά τον αντιτρομοκρατικό νόμο είναι κάτι που μας το είπαν και μας το ξαναείπαν. Έχουν γίνει καταχρήσεις, συνεχίζονται να γίνουν καταχρήσεις με άλλο την νομοθεσία αυτή. Ναι, ο κύριος Ντουντάρ βγήκε από τη φυλακή, πράγματι, αλλά πάνω από 90 μέρες έμεινε στη φυλακή. Είχαμε λοιπόν πολλές περιπτώσεις και ακαδημαϊκών οι οποίοι διώκονται από τον πρόεδρο επειδή ζήτησαν ειρήνη στο νοτιοανατολικό τμήμα της Τουρκίας. Καμία σχέση δηλαδή με την τρομοκρατία. Οπότε δεν μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους αφήσουμε στην τύχη τους, ούτε να αφήσουμε τους ανθρώπους να χάνουν τις δουλειές τους επειδή θέλουν ειρήνη στην ίδια τους τη χώρα. Έπειτα, ότι οι επικριτικές φωνές ε, ακούγονται, κλείνονται εφημερίδες κανάλια τηλεόρασης κλπ. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθούμε, γιατί εμείς θέλουμε η Τουρκία να προχωρήσει. Ήδη τα τελευταία 40 χρόνια είχε προχωρήσει η Τουρκία, είχε κάνει πρόοδους, οπότε δεν μπορεί τώρα να πηγαίνουμε πίσω. Η επικριτική από τον πρόεδρο ότι πρόκειται για τρομοκρατία. Και εσείς είπατε ότι πρέπει να υπάρχουν κοινοί ορισμοί για την ε, τρομοκρατία και την αντιμετώπιση της, αλλά για να επανέλθω και στο θέμα του συνήγορου του πολίτη. Ναι, υπάρχει στα χαρτιά. Στην πραγματικότητα όμως, οπότε ως κοινοβούλιο πρέπει όντως να κάνουμε και άλλα ταξίδια ε, τους επόμενους μήνες για να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα και, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν βασίζεται στο τι υπάρχει στα χαρτιά, αλλά στο ποια είναι η πραγματικότητα. Οι οργανώσεις γυναικών μας είπανε ότι απειλούνται, ότι εδώ και χρόνια δουλεύουν για τους θεσμούς, για τις ε, οργανώσεις υποστήριξης των γυναικών. Παρόλα αυτά τώρα ζουν με τον φόβο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν κοιτάει τι υπάρχει στην πραγματικότητα και όχι στη θεωρία. Ε, κύριε Χίκλ, ρωτήσατε διάφορα πράγματα. Αν τώρα πηγαίνουν κάποια κόμματα στην ακροδεξιά, το θέμα της εκπαίδευσης, ναι, έχει γίνει συζήτηση, τα ευρωπαϊκά μέσα το αναφέρουν, εμείς ασχολούμαστε με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένας πρόσφυγας είναι πρόσφυγας. Αν ένας πρόσφυγας χρειάζεται ένα καταφύγιο γιατί κινδυνεύει η ζωή του, τότε το θέμα δεν είναι του επίπεδου εκπαίδευσης. Εσείς αναφερθήκατε στην πρόσκληση της Μέρκελ. Αυτό είναι μια εθνικιστική προσέγγιση ακροδεξιά που ακούσαμε από συναδέρφους και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα βάζουμε την κυρία Μέρκελ, ότι εκείνη φταίει. Εντάξει, ήταν ηγετική φιγούρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως είναι στενόμυαλο όμως. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για την υποδοχή των προσφύγων και για το μέλλον, αλλάζοντας και το Δουβλίνο. Εμείς πρέπει να στηρίξουμε το λό της Τουρκίας και όχι να ασχολούμαστε μόνο με τον Ερδογάν. Εμείς συναντήσαμε ανθρώπους και από τον τύπο και ακαδημαϊκούς και από μη κυβερνητικέ οργανώσεις με ιδιαίτερο θάρρος. Αυτούς πρέπει να τους υποστηρίξουμε στο δρόμο που έχουν ακολουθήσει. Και να μην το περιορίζουμε σε αυτά που αναφέρατε εσείς, δεν θα τα επαναλάβω. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Λίτς. Θα συνεχίσουμε να συζητάμε για την Τουρκία της καλλιώς και τους επόμενους μήνες. Όσον αφορά την Υποβιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εννοείται ότι δεσμεύομαι απέναντί σας, ότι η Επιτροπή μας θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία. Αυτό που θεωρώ λάθος, όπως λέει και η κυρία Σχάκε, είναι να συνδέουμε τις διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της Τουρκίας με την προσφυγική κρίση. Αυτό δεν θα μας εμποδίσει να εκφράζουμε την άποψή μας για την διάκριση εξουσιών, ε, τα θέματα ισότητας ανδρών, γυναικών, μειονοτήτων, ελευθερίας έκφρασης κλπ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Πάλι στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί παραμένουμε. Πρόκειται για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη. Εδώ έχουμε μαζί μα τον κύριο Ρίκε Γκερέρο, ο οποίο προείδρευσε τι αντιπροσωπείε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διάσκεψη αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Ήταν η πρώτη ανθρωπιστική διάσκεψη που συγκλήθηκε ποτέ στην ιστορία. Τα Ηνωμένα Έθνη το αποφάσισαν και ο λόγος ήταν γιατί είμαστε σε μια στιγμή της ιστορίας ε, τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης ανά τον κόσμο. Είτε λόγω πολέμων, σειράξεων, είτε λόγω φυσικών ε, καταστροφών, πράγματα γνωστά. Ε, βέβαια που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή. Οι πρόσφυγες ανά το κόσμο σήμερα είναι πάνω από 60 εκατομμύρια. Δυστυχώς έχουμε αυτό το νούμερο. Μόλις αυτές τις κρίσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα εκατομμύριο έχει καλύψει. Ενώ το νούμερο των προσφύγων είναι πολύ μεγαλύτερο. Επίσης, η χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής κρίσης δεν είναι στα επίπεδα που θα έπρεπε. 40% λιγότερα είναι αυτά που δίνουμε. Πράγμα που σημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια οργανώσεις όπως των Ηνωμένων Εθνών για την ε, διατροφή αναγκάστηκαν σε κάποια σημεία του κόσμου να μην δίνουν πια τα τρόφιμα αυτά. Και επίσης πρέπει να αναθεωρήσουμε και την δομή της ανθρωπιστικής βοήθειας ανά τον κόσμο. Γι' αυτό συγκλήθηκε λοιπόν η διάσκεψη αυτή ακριβώς, γιατί είμαστε σε μια στιγμή της ιστορίας με πολύ οξύς ανθρωπιστικές κρίσεις. Επίσης, επειδή η δομή της απάντησής μας της ανθρωπιστικής δεν είναι ικανοποιητική. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Πολλοί παραβιάζουν τις ίδιες τις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας, τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Νόμο. Αυτή λοιπόν δεν ήταν μια διακυβερνητική διάσκεψη, ήταν μια διάσκεψη πολυμερής συμμετείχαν φυσικά και κυβερνήσεις από διάφορες χώρες, συμμετείχαν επίσης διεθνείς θεσμοί, μη κυβερνητικές οργανώσεις, χρηματοπιστωτικά χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, διάφοροι και γι' αυτό και υπήρχαν και προβλήματα, γιατί εννοείται πολύ θα θέλαμε όλοι να συμμετέχουν στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων. Από την άλλη μεριά όμως οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο τέλος είναι πολλές και διάφορες και δύσκολα ορατές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη δικιά της την πλευρά προετοιμάστηκε καλά για αυτή τη διάσκεψη. Υπήρξε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπήρξε έκθεση επίσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προετοίμασε αυτή τη διάσκεψη. Και εγώ ήμουν εισηγητή. Υπήρξαν δύο Ευρωπαϊκά Συμβούλια που εγκρίνανε συμπεράσματα προκειμένου να είναι φιλόδοξη διάσκεψη αυτή σε σχέση με τα αποτελέσματα που είχαμε στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα υπήρχε βέβαια ένα πρόβλημα που είχαμε και εμείς, δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Για τα Ηνωμένα Έθνη η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι ένα άγνωστο πολιτικό όν μη ξεκάθαρα προσδιορισμένο. Μερικές φορές αυτό ακούγεται και σε άλλες χώρες. Οι... Την μπερδεύουν τέλο πάντων την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρουν αν είναι η Λετωνία, αν είναι ποιος. Και αυτό ήταν μια δυναμία, όπως ξέρει πολύ καλά και η Έλενα Βαλενθιάνο, η πρόεδρός μας. Γιατί μέχρι την τελευταία στιγμή δεν γνωρίζαμε πραγματικά σε πόσες προσκλήσεις έπρεπε να ανταποκριθούμε. Τελικά το Κοινοβούλιο αποφάσισε για μια αντιπροσωπεία με μέλη από τρεις κοινοβουλευτικές επιτροπές, της ΔΕΒΕ, της ΔΡΟΑ και των γυναικών. Με 11 μέλη. Τελικά πήγαμε 5 γιατί ήταν αδύνατον να πάρουμε ουσιαστικές προσκλήσεις, προσκλήσεις που να μας επιτρέπουν να συμμετάσχουμε στις δραστηριότητες της διάσκεψης. Πρέπει εδώ να υπογραμμίσω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά μας έδωσε δύο προσκλήσεις οι οποίες ήταν για την Κομισιόν κανονικά προκειμένου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να είναι Παρόν με περισσότερους ευρωβουλευτές. Τέλος πάντων, είναι ενδιαφέρον να δείτε το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι ο βαθμός δεσμεύσεων που λήφθη στο τέλος. Πολύ light. Για να μην πω ότι και αυτές οι δεσμεύσεις είναι δύσκολα προσδιορίσιμες. Από πλευρά των Ηνωμένων Εθνών δεν υπήρξε πολιτική δήλωση που να συνυπογράφουν οι συμμετέχοντες, οι χώρε μέλη των Ηνωμένων Εθνών, για παράδειγμα. Υπήρξε μία δήλωση που προώθησαν οι Ηνωμένε Πολιτείε και που δέχτηκαν πολλές πλευρές, αλλά που δεν ήταν σε επίπεδο δεσμεύσεων, όπως απαιτούν οι συνθήκες. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά τις οικονομικές δεσμεύσεις, Μιλήσαμε για έναν μηχανισμό διαπραγμάτευσης που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Κρυσταλίνα Γεώργιεβα, εκείνη πρωτοστάτησε στην πρόταση αυτή. Στο μηχανισμό αυτόν δώσαμε το όνομα που δεν ξέρω αν είναι το πιο κατάλληλο, Great Bargain, μεγάλη διαπραγμάτευση, πώς να το πω. με τριαντατόσες υπογραφές που δεσμεύονται για διάφορα ζητήματα στο οποίο θα αναφερθώ. Δηλαδή, χρηματοδότηση για την ανθρωπιστική δράση που να διασφαλίζει προβλεψιμότητα. Δηλαδή να ξέρουμε τι έχουμε στη διάθεσή μας. Να προβλέπει επίσης ευελιξία στη χρήση των πόρων ε, αυτών και ευελιξία και στην αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών κρίσεων. Επίσης η δέσμευση για την προβλεψιμότητα σημαίνει ότι θα μπορούμε να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί. γιατί έτσι μπορεί να γίνει καλύτερο συντονισμός των πόρων. Υπήρξαν επίσης πολλές δηλώσεις επί της αρχής όσον αφορά την ανθρωπιστική δράση και την διεθνή ανθρωπιστική νομοθεσία, ε, προστασία από παραβιάσεις οι οποίες γίνονται σε πολλές περιπτώσεις των ανθρωπιστικών αρχών τα τελευταία χρόνια. Ακόμα ε, μιλήσαμε και για επιθέσεις σε βάρος ανθρωπιστικών υποδομών αυτό που μπορούμε να πούμε για τη διάσκεψη είναι ότι καθότι είναι η πρώτη, αποτελεί ένα σημείο κίνησης. Έτσι πρέπει να τη δούμε, σαν ένα πρώτο βήμα. Και πρέπει να δουλέψουμε ώστε το βήμα αυτό να γίνει δρόμος. Και ο δρόμος να γίνει αυτοκινητόδρομος. ώστε να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην ανθρωπιστική μας δράση. Ε, τρία σημεία. Το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Είναι το επόμενο βήμα όπου θα πρέπει να αποφασίσουμε για την υλοποίηση των όσων υπογράφηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Δεύτερο βήμα. Σε εμά εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει και εμείς να δουλέψουμε ώστε να συνδυάσουμε τις διεθνείς θεσμεύσεις που έχουν εγκριθεί 2015 και 2016 για την βιώσιμη ανάπτυξη, για την ε, χρηματοδότηση αντισαβέβα, κλιματική αλλαγή, διάσκεψη στο Παρίσι, η ανθρωπιστική αυτή εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα βάλουμε μαζί και να φτάσουμε έτσι στο τρίτο βήμα που θα είναι να ζητήσουμε από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο ένα σχέδιο δράσης προκειμένου όλες αυτές οι δεσμεύσεις από τις διάφορες διεθνείς διασκέψεις να αρχίσουν να υλοποιούνται. Προστασία από κινδύνους, αυτό που εγκρίναμε επίσης στην Ιαπωνία, στη Σαντάι πέρυσι. Σε όλα αυτά πρέπει να δώσουμε εμεί όθηση ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πρόγραμμα δράση, ένα σχέδιο δράση καθορίζοντα και ένα χρονοδιάγραμμα. Οπότε, για να καταλήξω, η διάσκεψη αυτή έλαβε χώρα την κατάλληλη στιγμή. Δεν ξέρω αν έγινε και μέσα στην καλύτερη δυνατόν ατμόσφαιρα γιατί υπήρχε και το θέμα της Τουρκίας από δίπλα. Αυτή τη φορά έγινε στην Κωνσταντινούπολη, θα μπορούσε να είχε γίνει αλλού και να μην είχαν συνδεθεί τα θέματα της ανθρωπιστικής βοήθειας με τα ζητήματα της Τουρκίας. Ήταν πάντως μια διάσκεψη πολυμερής με αδύναμες οικονομικές δεσμεύσεις, πολύ περιορισμένες και έχοντας υπόψη μας ότι η ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο απαιτεί περισσότερα. Όχι μόνο όσον αφορά τον τρόπο που τα αντιμετωπίζουμε, αλλά και την πρόληψη κυρίως, ότι πρέπει να τα προλαμβάνουμε όλα αυτά. Ε, το ξέρουμε, μπορεί να μην μπορούμε να προλάβουμε απαραίτητα έναν κυκλώνα, αλλά πάση περιπτώσει άλλα πράγματα που συμβαίνουν, οι σειράξεις, πόλεμοι. Όσες επιτροπές συμμετείχαν στην αντιπροσωπή αυτή, θα ετοιμάσουν κάποια έκθεση για τη συμμετοχή μας στη διάσκεψη. Αυτή είναι η πρώτη παρουσίαση στη δικιά μας την Επιτροπή τουλάχιστον. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Γκερέρο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Πολύ καλά τα εξήγησε ο συνάδελφος. Ωραία. Στη συνέχεια θα έχουμε μια επίσημη έκθεση για τις δραστηριότητές μας εκεί. Εγώ συμφωνώ πάντως με την ε, παρουσίαση του Ερίκη Γκερέρο. Ωραία, συνεπώς. Τελείωσε και αυτό το σημείο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκερέρο.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 ruego a todo el mundo que se sitúe. Καθίστε παρακαλώ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αρχίζουμε μία κρόση Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι στην καμπίνα 24 υπάρχει διερμηνία προς τα αραβικά. Οπότε, κύριε Γκερέρο, αν θέλετε να ακούσετε αραβικά, στο 24. Η 24 λοιπόν για τα αραβικά, κατά τα άλλα, ως συνήθως. Και αγγλικά, φυσικά και υπάρχουν και αγγλικά. Λοιπόν, έλεγα, ότι θα συζητήσουμε για ένα ζήτημα που ενδιαφέρει όλους ιδιαίτερο στην Υποπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρόκειται για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Μέση Ανατολή, κυρίως όμως πρόκειται για τις μειονότητες οι οποίες έχουν ε, παγιδευτεί στην Συρία, στο Ιράκ, Ντάς, Συρία, Υπάρχει επίση και δίωξη σε βάρος των χριστιανών στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε μαζί μας σήμερα πέντε προσκεκλημένους οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν την κατάσταση. Μια που γνωρίζουν πολύ καλά την κατάσταση σήμερα και έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Σαμ Άντρους πρώτα απ' όλα από το Arab Human Rights Academy. Ο Σαμ είναι προσωπικός βοηθός του εκτελεστικού διευθυντή της Ακαδημίας αυτής ακριβώς για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Αραβικής. Επίσης έχουμε μαζί μας την κυρία Σούντους Αμπάς που είναι πρόεδρος των ε, Τουρκμένων του Ιράκ στην Ευρώπη. Γεννήθηκε στο Κυρκούκ. Είναι μηχανικός έχει αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο του Αλτσαροντίν το 86. Προηγουμένως πήρε από το Πανεπιστήμιο του Greenwich δίπλωμα στην πληροφορική. Πήγε στην Αγγλία μετά από το δεύτερο πόλεμο του κόλπου και από το 2009 μέχρι το 2015 δούλεψε ως εκπρόσωπος του Ιρακινού μετόπου των Τουρκμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε μαζί μας και την κυρία Νάντια Μουράτ, η οποία είναι ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των Γεζιντής, που είναι μια θρησκευτική μειονότητα που διώκεται από το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος. Την απήγαγε τον Τας τον Αύγουστο του 2014, ακριβώς γιατί ήταν Γεζιντή. Πουλήθηκε σαν ε, σκλάβα, την βίασαν, αλλά κατάφερε να ξεφύγει από τους απαγωγείς της. Είναι λοιπόν μια ακτιβίστρια η οποία αφιερώνει τον χρόνο της για να προσφέρει μαρτυρίες όσον αφορά την κατάσταση του λαού της. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε σήμερα μαζί μας. 5 Ιανουαρίου του 2016 η Ρακινή κυβέρνηση την πρότεινε υποψήφια για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Έχουμε μαζί μας και τον πατέρα Ζιάντα Χιλάλ που είναι Σύριος Ισουίτης. Για έξι χρόνια οργάνωσε ανθρωπιστική βοήθεια για τους πρόσφυγες στα πλαίσια της υπηρεσίας των νησιτών για τους πρόσφυγες και διευθύνει ένα κοινωνικό κέντρο στη Χόμς που προσφέρει και ιατρική βοήθεια και ψυχολογική κλπ. Και έχουμε μαζί μας, για να δω θα το πω καλά, τον Εμμανουέλ Γιουκάνα πατέρα Μανουέλ Γιουκάνα, που είναι επικεφαλής των Ασσύριων Χριστιανών και επικεφαλής του Χριστιανικού Προγράμματος Βοήθειας στο Βόρειο Ιράκ. Όπως βλέπετε, όλοι αυτοί είναι άνθρωποι που προσφέρουν καθημερινά τη βοήθειά τους. Συγχρόνως όμως μπορούν και σε μας να μας παρουσιάσουν την κατάσταση για να καταλάβουμε καλύτερα τι συμβαίνει. Για να συνειδητοποιήσουμε καλύτερα τι γίνεται στην περιοχή. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι που ήρθατε εδώ. 12 λεπτό καθένας έχετε στη διάθεσή σας. Έχουμε χρόνο πάντως. Και θα αρχίσω δίνοντας το λόγο στον κύριο Σαμ Άντριους. Παρακαλώ κύριε Σαμ Άντριους, έχετε το λόγο. Το μικρόφωνο του ομιλητή είναι κλειστό. Το μικρόφωνο του ομιλητή είναι κλειστό. Τώρα ναι. Ξεκινώ λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σας. Έχουμε εκπροσώπους εννέα από τις εννέα ε, εκπροσώπους μενοτήτων. Θα ήθελα να σας δώσω μια σύντομη επισκόπηση αυτών των ε, ομάδων μενοτήτων του Ιράκ και κυρίως ε, των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στο Ιράκ σήμερα. Οι ομάδες που εκπροσωπώ είναι η Μαντέιν, 600 το πολύ, στο νότιο Ιράκ και τη Βαγδάτη. Το από, την, ε, από το 2003 έχουν εγκαταλείψει τη χώρα κατά το 90%. Έχουν εργαστεί παραδοσιακά ως ε, χρυσοχόοι, παίρνοντας χώρα τους. Έχουν υποστεί επιθέσεις, ε, και γενικότερα εκδήλωση βίας και μίσους. Έχουν αγκαστεί να εγκαταλείψουν τις ε, τους σε περιοχές όπου επικράτησε η ISIS, καθώς θεωρείται ότι δεν είναι ε, λαοί που πιστεύουν στη βίβλο, διώκονται. Η θρησκεία τους στηρίζεται στην ύπαρξη καθαρού τρεχό, τρεχούμενου νερού και όπου δεν μπορούν να το βρουν δεν είναι στη θέση να παρακολουθήσουν τις παραδόσεις τους. Είναι υπό την προστασία της UNESCO και προσπαθούν να επιβιώσουν. Το πρόβλημα επιδεινώνεται με, την, με τους εκτοπισμούς, τις οικονομικές πιέσεις και τις διακρίσεις. Οι Μαντέν έχουν επίσης τον κίνδυνο να εξαφανιστούν ως κοινότητα λόγω των εκτοπισμών αυτών. Μόνο δια της γέννησης μπορεί κανείς να διαιωνίσει αυτήν την κοινότητα. Έχουμε λοιπόν τους Παλαιστίνιους υπό την ε, διοίκηση του Ιράκ που χαρακτηρίστηκαν ως υποστηρικτές του Σαντάμ Χουσένου το 2030, υφίστανται πολλές ε, διώξεις επιθέσεις, ε, δυσφημίσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, βασανιστήρια, δολοφονίες και πολλοί έχουν αναγκαστεί να διαφύγουν στα εξωτερικά κράτη, Συρία και η Ορδανία. Θεωρείται μάλιστα ότι το Ιρακινό Υπουργείο των Εσωτερικών είναι συνένοχος σε αυτές τις επιθέσεις εις των Παλαιστινίων, οι οποίοι και λόγω απουσίας ε, εντολής της Ούγγρα για το Ιράκ δεν έχουν καμία προστασία εκεί και δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Η Σαμπάκ επίσης, 250.000, κυρίως στο βορρά. Μουσουλμάνοι Σι, περισσότεροι, δεν θεωρούνται ούτε Άραβες ούτε Κούρδοι. Ζουν όμως σε μια διφυλονικού περιοχή και ω εκ τούτου έχουν πέσει θύματα διαφορών πολιτικών που ανατρέπουν τις δημογραφικές ισορροπίες. Η κυβέρνηση ε, το καθεστώς του, του Μπαφ είχε προσπαθήσει να τους ενσωματώνει σε ένα πρόγραμμα εξαραπισμού. Από το 2003 έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.300. Είναι πολλές οι πιέσεις που υφίστανται όταν βρίσκονται σε στρατόπεδα εσωτερικά εκτοπιστέντων να ταυτοποιηθούν ως Κούρδοι. Έχουν υποστεί πολλές δίωξεις από, το Ίσις λόγω της ε, απόρριψης από πλευράς τους της ερμηνείας του σαλαφικού τύπου, αγαβιστικου τύπου του Ισλάμ. Η Μπαχάοι γύρω στους χίλιους, δεν υπάρχουν πιστές ε, στατιστικές για αυτούς, ήταν παράνομη θρησκεία τους υπό το καθεστώς του Μπαθ. Δεν μπορούσαν να γράψουν τη θρησκεία Μπαχάη στις ταυτότητές τους από την απαγόρευση αυτής της καταχώρησης του 2007. Πολλοί προσπάθησαν να καταγράψουν τη θρησκεία τους, γιατί πριν ε, δηλώνονταν ως μουσουλμάνοι μόνο. Αλλά ο νόμος παριθμών 105 δεν ε, ανακλήθη ποτέ και έτσι δεν μπορούν να έχουν τα σχετικά έγγραφα ταυτότητας. Οι Ρωμά από 50 200.000 ζουν κυρίως σε απομονωμένα χωριά στο Νότιο Ιράκ στη ε, περιχώρα της Βαγδάτης, της Βασόρας και της Μοσούλης. Δεν έχουν βασικές υπηρεσίες, ε, τους ε, στοχεύει το ίσως και λόγω των παραδοσιακών τους ενασχολήσεων ως ανθρώπων της αναψυχής μουσικών, χορευτών κτλ. Η Κούρδοι Φεϊλοί, 1,5 εκατομμύριο επίσης ΣΥ, έχουν αντιμετωπίσει σιήτες, έχουν επίσης αντιμετωπίσει πολλές διώξεις. Το 2012 είχε υπολογιστεί ότι 120.000 ήταν οι απάτριδες, εκ των οποίων μεγάλο ποσοστό ήταν φίλοι. Οι μαύροι Ιρακινοί όπως ονομάζονται, 1,5-2 εκατομμύρια, κυρίως στο νότιο Ιράκ, από και στην περιοχή της Βασόρας, αλλά και στο βορρά, στη Ραμπέα, κοντά στη Μοσούλη, ε, με ποσοστά ανεργίας μέχρι και 80% και απουσία παροχής των βασικών υπηρεσιών, πολλές διακρίσεις εις βάρους τους, εκτεταμένος κοινωνικός αποκλεισμός. Μπορεί να, υπάρχει, να είναι μεγάλο το μέγεθος της κοινότητάς τους, αλλά κανένας τους δεν έχει αναλάβει πολιτικά καθήκοντα. Υπήρξε το ελεύθερο Ιρακινό κίνημα με εκστρατείε για τα δικαιώματα των μαύρων Ιρακινών, αλλά ο ιδιαίτερη του δολοφονήθηκε το 2013. Η Κακάη επίσης 200.000 ε, κοντά στις περιοχές του Κυρκούκ, ε, κυρίως Κούρδοι, με μια θρησκευτική παράδοση που συνιστά μείγμα ζωροαστρισμού και Ισλάμ. Πολλές φορές έχουν ε, πέσει θύματα συστηματικών διακρίσεων, καταχρήσεων, απαγωγών, δολοφονιών. Του στοχεύει το ίσως, θεωρεί ότι είναι αποστάτες δηλαδή, γιατί και η θρησκεία τους είναι απόκριφη και δεν είναι εύκολο να τους προσεγγίσουν και γι' αυτό λόγο οι ανθρωπιστικές οργανώσεις. Οι Ιρακινοί Εβραίοι με μονοψήφιο ή διψήφιο το πολυνούμερο που είναι δύσκολο να υπολογιστεί. Πριν από τις ε, διώξεις τη δεκαετία του 50 υπήρχαν 120.000 Εβραίοι στο Ιράκ. Τώρα δεν μπορούν να διαφυλάξουν την περιουσία τους. Έχουν πολύ λίγα δικαιώματα, κινδυνεύει η παράδοσή τους στο Ιράκ. Έχουμε εκπρόσωπο των Εβραίων στην κεντρική δίκη από το 2015, αλλά δεν μπορούν να διαφυλάξουν βασικά πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα. Η ανάδειξη της ε, οργανώσης ίσης ε, επέτεινε τα προβλήματα αυτά, καθώς διακρίσεις και η βία είναι κύρια χαρακτηριστικά του προγραμματός, αλλά ήδη βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση αυτές οι κοινότητες, ήδη αυτές που βρίσκονται στο Βόρειο Ιράκ, Πολλές φορές εγκλήματα εις βάρος των κοινωτών αυτών τα αγνοεί η αστυνομία και λόγω του διαφθοράς αλλά και λόγω διακρίσεων. Γενικά βλέπουμε ότι ο χώρος της ταυτότητας, της αθηματικής ταυτότητας μέσα στην Ιρακινή κοινότητα έχει συσταλεί λόγω του πολέμου με το ίσης. Ε, δεν επιτρέπεται να κάνεις διαφορετικός δηλαδή και στενεύουν τα όρια του τι σημαίνει να κάνεις Ιρακινός, Κούρδη και άλλοι ε, δεν μπορούν να μιλήσουν πλέον, δεν μπορούν να έχουν χώρο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Επιτροπή και Τηλεπικοινωνιών και μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που τώρα προσπαθεί να κατασυγάσει οποιαδήποτε επίκριση εις βάρος της ε, κυβέρνησης, των δυνάμεων που υποστηρίζουν την κυβέρνηση, ε, ενώνει έχουν περισσότερο το πρόβλημα. Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι χαρακτηριστικό, μια χαρακτηριστική εμπειρία των κοινωνιών αυτών, των κοινωτήτων αυτών δεν υπάρχουν πλατφόρμες πολιτικές για κινητοποίηση και διεκδίκηση δικαιωμάτων. Η βία που υφίστανται ιδιαίτερα μπορεί να παραβλάψει τις κοινότητες που έχουν τόσο μικρό αριθμό μελών και για λόγους γεωγραφικής συγκέντρωσης ή επειδή είναι αποκομμένες από την υπόλοιπη χώρα, από τον υπόλοιπο πληθυσμό, οι απώλειες τους θα είναι καταστροφικές όχι μόνο αριθμητικά αλλά και σε επίπεδο πολιτικού και κοινωνικού δικτύου. Κάποια μέλη των κοινοτήτων που έχουν μεγαλύτερε διαστάσει μπορούν να μετακινηθούν σε άλλε περιοχέ και εάν έχουν εκεί ομοεθνεί να εξασφαλίσουν υποστήριξη, ενώ αυτοί που ανήκουν σε μικρότερε κοινότητε δεν έχουν κανένα ασφαλέ μέρο να καταφύγουν. Είναι περίπλοκη κατάσταση λοιπόν, με ιδιαίτερε συνθήκε, Η οικονομική βοήθεια με ένα πακέτο 850 δολαρίων για την καταγραφή των ιστορικά εκτοπιστέντων είχε διατεθεί αλλά δεν είχαν τα δελτία ταυτότητας ε, κοινότητες όπως Παλαιστίνη, Μπαχάη, Φίλοι και ήταν πολύ δύσκολο να τους προσφερθεί υποστήριξη. Τα προβλήματα λοιπόν δεν φαίνεται να λαμβάνουν υψηλό βαθμό προτεραιότητας για τις αρχές και αντίθετα χρησιμοποιούνται ε, τα στοιχεία ορισμένες φορές των εσωτερικών σεκτοπιστέντων ανεξαρτήτως της προέλευσης και της ε, κοινότητας στην οποία ανήκουν προκειμένου να ε, υποστηριχθούν δημογραφικά επιχειρήματα. Δεν υπάρχουν πόροι και στήριξη, ειδικότερα για τις μικρές ομάδες. Δυστυχώς δεν έχω και το χρόνο για να καλύψω την μεγάλη πληθώρα των διαφορών αυτών των ομάδων, τα περίπλοκα χαρακτηριστικά της σύγκρουσης. Και έτσι πολλά δυστυχώς θα πρέπει να τα παραλείψω. Οι γυναίκες, παραδείγματι, που υποφέρουν, γυναίκες αυτών των μικρών μειονοτικών ομάδων υποφέρουν ιδιαίτερη βία, πολύ συχνά σεξουαλικές ε, επιθέσεις, βιασμού ακόμα και δολοφονίες προκειμένου να αποστελεί και ένα μήνυμα ή να, τους τους να τις αποστερήσουν και από την ε, ανθρώπινη τους υπόσταση ακόμη. Μπορεί να μην έχουν ασφαλή δίκτυα κοινωνικά για να το στηρίξουν οι κοινότητές τους, εάν αυτές φωνευτούν ή αν εκτοπιστούν. Και βλέπουμε ότι πολύ συχνά η ζημία αναπτύσσεται σε πολλαπλά επίπεδα και για να εξασφαλιστούν ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράκ χρειάζεται μια πιο περίπλοκη προσέγγιση, δεν μπορούμε να έχουμε μια μόνο κόμματη, μόνο διάσταση προσφορά λύσεων. Πρέπει να ακούσουμε τους ανθρώπους αυτούς, να αντιλημιληθούμε τα προβλήματα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά. Σας ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Άντριους, για τον τρόπο με τον οποίο συνοψίσατε το θέμα. Ευχαριστώ. Η κυρία Σούντου Σαμπάς έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, καλησπέρα σας. Εγώ σήμερα εκπροσωπώ τους ε, τουρκομάνους ε, του Ιράκ. Ε, είναι η τρίτη εθνοτική ομάδα στο Ιράκ. Είναι περίπου 3 εκατομμύρια άτομα, 13% του Ιρακινού πληθυσμού. Κυρίως στη Μοζούλη, στο Καρκούκο, στο Σαλαντίν και στη Διάλα ε, η, το Κυρκούκ ε, θεωρείται η πρωτεύουσα για τους Τουρκομάνους, όμως ε, η κεντρική κυβέρνηση στη Βαγδάτη και η κουρδική περιφερειακή κυβέρνηση συνεχώς συγκρούονται προκειμένου να διεκδικήσουν αυτήν την ε, πόλη, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πάρα πολλές κατασχέσεις γίνονταν ε, από τον Σαντάν Χουσεΐν τότε και μετά το 2003 ε, από την κεντρική κυβέρνηση, απλώς και μόνο για να γίνει μια δημοκρατική αλλαγή στην περιοχή. Ε, ήταν πάντοτε ο πληθυσμός αρκετά, ε, παρουσίαζε μεγάλη ποικιλία, υπήρχαν χριστιανοί, υπήρχαν ε, τουρκομάνοι και οι τουρκομάνοι πάντοτε ήταν αντικείμενο καταπίεσης και τους πίεζαν να λένε ότι είναι Κούρδοι πάντοτε ήταν θύματα προσπάθειας ε, ομογενειοποίησης, ε, ήταν αντικείμενα εθνοκάθαρσης και δεν είχαν ποτέ το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, αυτονομία ή οποιοδήποτε, οποιοδήποτε ρόλο ε, στα, στον, βίο, στον κοινωνικό και πολιτικό βίο του κράτους. Κάτι το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται και σήμερα. Αυτό ξεκίνησε κατά το καθεστώς του ΠΑΘ μετά από την πτώση του καθεστώτος του Χουσέιν το 2003. Όλοι οι Ιρακινοί είχαν ε, μεγάλες προσδοκίες ότι ε, θα άλλαζαν τα πράγματα μετά από την κυβέρνηση που ανέλαβε τον Απρίλιο του 2003 οι Τουρκομάνοι περίμεναν δικαιοσύνη, δημοκρατία, ποιότητα, ισότητα, δικαιοσύνη και το τέλος των διακρίσεων, το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και το τέλος της βίας. Όμως δυστυχώς συνέβη το αντίθετο. Από το 2003 ε, άρχισαν να γίνονται βομβιστικές επιθέσεις κατά των Τουρκομάνων, απαγωγές, δολοφονίες ε, σε όλες τις περιοχές όπου ζουν οι Τουρκομάνοι. Εκτίθενται σε τεράστιο βαθμό ε, σε συλλήψεις, ε, πάρα πολλοί αγνοούμενοι μάλιστα ε, είναι τουρκομάνοι και 95% των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Ιράκ είχαν ως στόχο τους τουρκομάνους, δικηγόροι, γιατροί έχουν λάβει απειλές για ενδεχόμενη απαγωγή τους ή δολοφονία τους. Περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια έχουν πληρωθεί σε λίτρα προς τους απαγωγείς. Οι γειτονιές των Τουρκομάνων δεν έχουν καμία προστασία παρά το γεγονός ότι υπάρχει ε, ασφάλεια που προστατεύει άλλες περιοχές οποίες δεν διαμένουν Τουρκομάνοι. Ε, οι περισσότερες μειονότητες έχουν μία παρουσία στις δυνάμεις ασφαλείας, όμως οι Τουρκομάνοι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό και δεν συμμετέχουν καθόλου στην διαδικασία λήψης αποφάσεων στον Ιρακινό στρατό, κάτι το οποίο τους έχει καταστήσει πιο ευάλωτους σε επιθέσεις και τρομοκρατία. Ε, κάθε περιοχή όπου ζουν οι Τουρκομάνοι ε, έχουν ε, αποτελέσει, έχει αποτελέσει αντικείμενο τρομοκρατικής επίθεσης από το 2003 μέχρι το 2013 έχουν ε, ζητηθεί, έχει ζητηθεί ύπαρξη μέτρων για την ε, ενίσχυση των τουρκομάνων και τη διαφύλαξη της ασφάλειάς τους, όμως δεν έχει ληφθεί καμία απολύτως απόφαση. Η ε, κουρδική κυβέρνηση εξακολουθεί να αντιστέκεται ε, στην ύπαρξη ασφάλειας στις περιοχές αυτές ε, με αποτέλεσμα να υπάρχει διάκριση και βία κατά των Τουρκομάνων στις περιοχές όπου διανέμουν. Μετά που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στο Ιράκ και άρχισαν βέβαια με στόχο τις ε, περισσότερο ευάλωτες ομάδες όπως τους Γεζίδιδες, τους Τουρκομάνους και τους Χριστιανούς δεν έχουν τις δικές τους δυνάμεις ασφαλείας για να τους προστατεύσουν οι ομάδες αυτές. Στις 15 Ιουνίου του 2014 οι αγωνιστές ε, του ISIS πήραν ε, την Τέλαφορ που είναι ε, μια βασική πόλη στην οποία διαμένουν Τουρκομάνοι. Πάνω από 350.000 Τουρκομάνοι έφυγαν από την πόλη αυτή. Το ISIS απήγαγε τουλάχιστον 150 παιδιά και πάρα πολλές γυναίκες και τους χρησιμοποίησαν με διαφορετικούς σκοπούς, ε, βιασμοί, δουλεία. Ε, πάρα πολλές ε, οικογένειες Τουρκομάνων έπρεπε να φύγουν από τη Μοζούλη και να διαφύγουν σε γειτονικέ περιοχές. Πάνω από 70 παιδιά ε, έχασαν τη ζωή τους επειδή δεν υπήρχε νερό και ήταν πολύ ψηλές οι θερμοκρασίες την ημέρα που έφυγαν από την Τελαφόρ τον ε, Ιούνιο του 2014 έγινε μια τρομοκρατική επίθεση με απαγωγή, ε, βιασμό και δολοφονίες παιδιών και γυναικών. Ε, οι περισσότερες περιοχές καταστρέφονται ολοσχερός. 700 Τουρκομάνοι δολοφονήθηκαν, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες και χιλιάδες οικογένειες έφυγαν από την Μπασίρ. Ε, οι γυναίκες ε, πολλές φορές δολοφονήθηκαν και κρεμάστηκαν τα κεφάλια τους ε, στα στις κολόνες ηλεκτροδότησης. Πρόκειται για μια ομάδα η οποία αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα επίθεσης και τρομοθετικών επιθέσεων και δεν υπάρχει καμία ασφάλεια. Ε, όταν γίνονται οι επιθέσεις, οι άνθρωποι αδιακρίτως δολοφονούνται, ηλικιωμένοι γυναίκες, μικρά παιδιά, κάποιοι καταφέρουν να φύγουν αφήνοντας πίσω τους, τους πιο ευάλωτους οι οποίοι δολοφονούνται ή βιάζονται, ε, ενώ όλο τους το βιός καταστρέφεται. Ε, μία ακόμη ε, πόλη Τουρκομάνων ε, ήταν υποπολιορχία έξι ολόκληρες ημέρες τέλη Ιουλίου και αρχές Αυγούστου 2014 υπό απάνθρωπες συνθήκες χωρίς να υπάρχει ηλεκτροδότηση, χωρίς να, υπάρχει καθόλου, να υπάρχουν καθόλου τρόφιμα ε, πάνω από 50 ε, παιδιά, 10 νεογέννητα έχασαν τη ζωή τους ε, επειδή δεν υπήρχαν τρόφιμα. Πάνω από 100 άτομα χάθηκαν λόγω της πολιορκίας και των καθημερινών επιθέσεων. Στις 10 Μαρτίου 2016 ε, το ISIS ε, επιτέθηκε στην Τάζα που είναι μια μικρή πόλη τουρκομάνων ε, νότια των του Κυρκούκ. Πάνω από 3.000 Τουρκομάνοι χάθηκαν ή βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η επίθεση έγινε με χημικά όπλα δεν έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες κατά των Τουρκομάνων από το 2003, αλλά έχει επιδεινωθεί κατά τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια πάνω από 150.000 άτομα, από 1.500 άτομα ε, έχουν, ε, ε, πάνω από έχουν αποκεφαλιστεί και χιλιάδες οικογένειες πρέπει να φύγουν από τις χώρες, από τις περιοχές στις οποίες μένουν προς την Βαγδάτη για παράδειγμα όπου η ζωή τους εξακολουθεί να βρίσκεται σε κίνδυνο. ανάμεσα στο, μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου του 2016 Κούρδοι Πεσμεργά μαζί με το ΠΚΚ επιτέθηκαν ε, με ε, βαρύ οπλισμό ε, σε τουρκομάνους και κατέστρεψαν τα σπίτια τους και μπορώ να ολοκληρώσω την ομιλία μου λέγοντας ότι οι πιο πρόσφατες επιθέσεις κατά των τουρκομάνων δεν είναι κάτι το καινούριο, είναι το αποτέλεσμα δεκάδων χρόνων εκφοβισμού από τους Κούρδους με σκοπό να τους ε, μετατοπίσουν από τις περιοχές οι οποίες μένουν εδώ και αιώνες. Γιατί εμείς είμαστε Τουρκομάνοι που ζούσαμε σε συγκεκριμένες περιοχές ε, ε, όταν οι Ιρακινές περιοχές δεν είχαν καθόλου δυνάμεις ε, ασφαλείας, κυρίως οι Πεσμεργά προσπάθησαν να ε, αναλάβουν την ηγεσία των χωρών αυτών, με αποτέλεσμα οι Τουρκομάνοι να μείνουν απολύτως ε, εκτεθειμένοι. Υποχρεώθηκαν να φύγουν περίπου 600.000 Τουρκομένοι από τις περιοχές όπου έμεναν, δεν έχουν στέγαση, δεν έχουν ιατρική περίθαλψη, δεν υπάρχει ιατρική φροντίδα είδα οι περισσότερες εκτοπιστήσεις οικογένειες δεν έχουν ε, καθόλου χαρτιά, δεν έχουν καθόλου ε, ταυτότητες και εξαρτώνται από χαρτιά που τους δίνουν ε, φιλανθρωπικές οργανώσεις, συνταξιο, συνταξιούχοι, ηλικιωμένοι, άνθρωποι με αναπηρίε, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επηρεάστηκαν περισσότερο. Ε, μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης, των Κούρδων, του ΠΚΚ και του ΆΙΖΙΣ είναι παγιδευμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Η διεθνής κοινότητα ε, αγνοεί ε, την κατάσταση αυτή που πλήττει τους Τουρκομάνους εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν κάνει τα απαραίτητα ώστε να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ενταχθούν, ώστε να υπάρχει σταθερότητα και δικαιοσύνη στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Η Νάντια Μου έχει τώρα το λόγο, λέει η πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω την ε, Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόσκλησή της σήμερα. Οι μειονότητες οι θρησκευτικές δηλαδή μειονότητες, εδώ και πολύ καιρό αποτελούν αντικείμενο μελέτης όχι μόνο εξαιτία του λεγόμενου Ισλαμικού <coughs> κράτους, αλλά είναι κάτι που έχει να κάνει με την ίδια την ιστορία της περιοχής. Είχαμε την Αραβική Άνοιξη, η οποία άλλαξε την κατάσταση εκεί, στο Ιράκ, στην Ιεμένη, στη Λιβύη για παράδειγμα. Ίσως στην Αίγυπτο και την Τινησία τα πράγματα να ήταν κάπως διαφορετικά, γιατί οι χώρες αυτές κατάφεραν να εγκαθιδρύσουν ένα δημοκρατικό σύστημα. Εκεί όμως όπου υπήρχαν θρησκευτικές μειονότητες η κατάσταση δεν ήταν εύκολη. Οι μειονότητες αυτές αφορούν εκατοντάδες, ή μάλλον παλιότερα ήταν εκατοντάδες χιλιάδες, τώρα είναι μερικές εκατοντάδες ψυχές που αποτέλεσαν αντικείμενο συστηματικής δίωξης τα τελευταία χρόνια. Στην Τουρκία οι γυζιδιά θεωρούνται άπιστοι. Στο Ιράκ επίσης διώκονται για θρησκευτικούς καθαρολόγους. Οι διώξει αυτές γίνονται με διαφορετικούς τρόπους. Εγώ εδώ θέλω να αναφερθώ στις διάφορες μειότητε της περιοχή και όχι μόνο του Γεζίδη, γιατί εγώ δεν βλέπω διαφορά ανάμεσα στη μία και την άλλη μειονότητα. Ένας άνθρωπος είναι άνθρωπος, όπου και αν βρίσκεται. Η γη είναι για όλους μας. Οι ανθρωπιστικέ αξίε είναι αυτέ οι οποίε μα ενώνουν όλου. Αυτές οι αξίες μας αναγκάζουν να αντιμετωπίζουμε τον άνθρωπο με τον ίδιο τρόπο από ποια φυλή και αν προέρχεται, από ποιο έθνος ή θρησκεία. Θα μιλήσουν άλλοι για επιμέρους τμήματα του μοσαϊκού αυτού. Εγώ θα επικεντρωθώ στους Γεζιντή. Πρέπει να ξέρετε ότι όλες οι μειονότητες στη Συρία και στο Ιράκ διώχτηκαν με το χειρότερο δυνατόν τρόπο οι σαμπάκι, οι σίτες ε, έχουν διωχθεί σε ολόκληρη την περιοχή της Συρίας. Απαλατριώθηκαν ε, οι υγιές τους, τους κατάσκεσαν τα καθά τους. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δικαιώσουμε τους ανθρώπους αυτούς Υπάρχει κόσμος που αναγκάστηκε να φύγει εξαιτία του πολέμου ή που έχασε και τη ζωή του, αλλά υπάρχουν και αυτοί που διώκονται ακριβώς επειδή ανήκουν σε μια θρησκευτική μειονότητα. Αυτό συνέβη με τους Γεζεντή ιδιαίτερα. Τους επιτρέπουν ή να ληξοπιστήσουν Ισλάμ ή να τους σκοτώσουν. Άλλες ε, μειονότητες είχαν κάποιες διαφορετικές δυνατότητες να πληρώσουν, για παράδειγμα, Όμως στις μουσουλμανικές κοινότητες πιστεύουν ότι οι Γιαζεντοί είναι άπιστοι, ότι είναι κακοί, δεν αναφέρονται καν στο Κοράνι και τέτοιες λαθασμένες πληροφορίες έχουν σαν αποτέλεσμα οι Γιαζεντοί να είναι αυτοί οι οποίοι διώκονται περισσότερο από τους τρομοκράτες. Οι γυναίκες τους βιάστηκαν, συλλαμβάνονται εξαιτίας της θρησκείας τους και μόνο. 74 διαφορετικές σφαγές έλαβαν ε, χώρα κατά τη διάρκεια της ιστορίας τους στη Σιντζάρ. 5.000 γιαζιντοί σκοτώθηκαν ε, στις 3 Αυγούστου 2014. 6.000 γυναίκες και παιδιά ε, έγιναν σκλάβοι. Καταστράφηκαν θρησκευτικές περιοχές, και πάνω από 80% της κοινότητας αυτής αναγκάστηκε να εκτοπιστεί χωρίς να έχουν τα βασικά εκπαίδευση, υγεία ή άλλες υπηρεσίες από το 2014 μέχρι τώρα. Υπάρχει λοιπόν μια γενοκτονία σε βάρος των Γιαζιντή που συνεχίζεται. Πέρασε 1,5 χρόνος. Παρόλα αυτά βρίσκονται κρατούμενοι 3.300 γυναίκες και παιδιά και κατά την κράτησή τους αυτοί είναι θύματα τεράστιων εγκλημάτων, ψυχολογικών μεταξύ άλλων. Και φυσικά η τάση είναι υπεύθυνη. Ο ανιψιός μου, 13 χρονών, βρίσκεται υπό πλήση εγκεφάλου. Τον έχουν πείσει ότι η οικογένειά του είναι η άπιστη. Υπάρχουν χιλιάδες χείρες, ορφανά και όπως σας είπα δεν έχουν καμία βοήθεια, καμία προστασία και δεν ξέρουν τίποτα για τις οικογένειές τους Στην ε, Φελούζα και στην Ράκα σήμερα το ξέρετε ότι οι γυναίκες και τα παιδιά μας χρησιμοποιούνται σαν ανθρώπινες ασπίδες. Δεν μπορούν να φύγουν γιατί τους προορίζουν για το θάνατο. Γιατί λοιπόν να θυσιάζονται αυτοί οι αθώοι. Γιατί να σκοτώνονται με τέτοιο τρόπο. Το έγκλημα της γενοκτονίας συνεχίζεται σε βάρος των ανθρώπων αυτών, ακόμα και σήμερα. Ψυχολογικά η κατάστασή τους είναι πολύ άσχημη, αλλά και η ζωή τους ίδια. Τους ε, πήραν, όπως σας είπα, τη γη τους, τα υπάρχοντά τους, πράγματα τα οποία τελικά δεν έχετε η διεθνής κοινότητα. 60% στη Σίντσα ελευθερώθηκαν, αλλά δυστυχώς η Ντάς τα έχει καταστρέψει όλα στην περιοχή. Οι γιαζιδοί δεν μπορούν να ζήσουν εκεί από όπου έχουν, έχει περάσει η 80% δηλαδή των γιαζιδοί αναγκάζονται να ζήσουν σε καταβλισμούς κάτω από τραγικές συνθήκες μέχρι να βρεθεί μια πολιτική και στρατιωτική λύση στην περιοχή. Στις ελευθερωμένες ε, περιοχές βρέθηκαν 35 ε, κινητάφοι όπου βρέθηκαν τα πτώματα 80 γυναικών για ζητή. Μεταξύ αυτών και η δικιά μου η μητέρα. Όλα αυτά βέβαια βγαίνουν στο φως κάτω από την διαφορία θα έλεγα της ε, διεθνούς κοινότητας και δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα. Γι' αυτό ακριβώς και κάνω έκκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από εδώ να έρθει σε επαφή με τις κυβερνήσεις ώστε να γίνει κάτι ώστε να αναγνωριστεί η γενοκτονία σε βάρος της κοινότητάς μας. Στη Σίντζα αλλά και στο χωριό μου, στο Κόχο, 700 άντρες δολοφονήθηκαν στις 15 Αυγούστου που μας πέρασε. Η ΝΤΑΣ βέβαια είναι περήφανη για τα εγκλήματα αυτά σε βάρος των Γιαζιντή. Μάλιστα δημοσιεύει και βίντεο ή φωτογραφίες όπου αναγνωρίζουν ανοιχτά τα εγκλήματά τους αυτά. Ότι έχουν ε, δηλαδή ε, συλλάβει και έχουν κάνει σκλάβους, γυναίκες και παιδιά. Είναι πράγματα τα οποία τους επιτρέπει ο δικός τους ο νόμος. Εμείς θέλουμε το έγκλημα αυτό της γενοκτονίας να αναγνωριστεί. Δυστυχώς δεν έχει γίνει αυτό μέχρι σήμερα. Εμείς έχουμε καταθέσει επαρκείς αποδείξεις για να ξεκινήσει μια διεθνής έρευνα. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές δυνατότητες για να παρουσιάσει κανείς ε, τα γεγονότα αυτά και να τα υποβάλει στο Διεθνής Ποινικό Δικαστήριο. Θέλουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας βοηθήσει σε αυτό. Η δικαιοσύνη είναι ο μόνος δρόμος που θα βοηθήσει να φτάσουμε στην ειρήνη. Έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε τους Γεζεντή αλλά και άλλους ώστε να μπορέσουν να βρουν την ειρήνη στη γη τους. Αν ο κόσμος δεν είναι σε θέση να κυριαρχείται από τη δικαιοσύνη, τότε τι θα κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί να φεύγουν από τη γη τους και να μην μπορούν να βρουν έναν χώρο ειρήνης κάπου αλλού, δηλαδή που να είναι ασφαλής. Κάπου 2587 για ζητή, γυναίκες και παιδιά κυρίως κατάφεραν να το σκάσουν από τον ΤΑΣ και χρειάζονται ψυχολογική βοήθεια, ιδιαίτερη ψυχολογική βοήθεια, γιατί ζουν κάτω από φρικτές συνθήκες στους καταβλισμούς του Κουρδιστάν, στο Ιράκ. Η Γάδη Βούρτεβούργη στην Γερμανία έχει ήδη υποδεχτεί 1.100 επιζήσαντες από αυτούς. Κι εγώ ίδια βρέθηκα εκεί. Παρ' αυτά παραμένουν 1.600 γυναίκες και παιδιά που παραμένουν στους καταβλισμούς και που χρειάζονται και αυτή την ίδια ψυχολογική βοήθεια. Σήμερα οι εξτρεμιστές τα βάζουνε με τους Γεζιντή όχι μόνο στη, στο Ιράκ, ε, στη Συρία αλλά και στην Τουρκία και στην Ελλάδα στους καταβλισμούς και στη Γερμανία ακόμα. Η τύχη δηλαδή σήμερα το Γεζιντή είναι η τύχη που επιφέλεξε το Τρίτο Ράιχ στους Εβραίους. Το ίδιο ακριβώς όπως με τους μαύρους της Αμερικής πριν από το 1960. Στο Ιράκ και στη Συρία λοιπόν οι μειονότητες κινδυνεύουν. Πρέπει να βρούμε λύσεις για να τους ανακουφίσουμε. Και για να συνοψίσω, η λύση είναι εξή. να ελευθερώσουμε τη γη, το έδαφος, να διασφαλίσουμε στρατιωτικά την ασφάλεια και τη διεθνή προστασία για τον κόσμο εκεί. Ζητάω επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει ένα ειδικό ταμείο για την ανοικοδόμηση του Σιντζάρ και άλλων περιοχών των Γιαζιντή και αυτό υπό διεθνή εποπτεία. Συζητώ επίσης να μας βοηθήσετε να ετοιμάσουμε το φάκελό μας για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ώστε να βασιλεύσει η ειρήνη. Να επηρεάσετε κι εσείς τα πράγματα. Τέλος, ζητάω να επιτρέψουμε στους μετανάστες να φτάσουν 7.000 Γιαζιντοί στην Ελλάδα και την Τουρκία. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Πάτερ Ζιάντι Λάλα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Θα μιλήσω γαλλικά. Δεν γνώριζα ότι θα μπορούσα να μιλήσω αραβικά. Από την απαρχή της κρίσης η Εκκλησία έζησε και υπέστη όλα αυτά που έχουν ζήσει και υποστεί οι Σύριοι πολίτες, ε, δίνα, πόνο, ακόμα και διχασμό. Παρ' όλα αυτά και παρά τα δικά της ε, δίνα και όσο ότι έχει γίνει πολύ πιο ευάλωτη, δεν εγκατέλειψε ποτέ το καθήκον της στην ε, ανθρώπινη και ανθρωπιστική της αποστολή για όλους τους Σύρους. Ξέρετε ότι έχουμε δύο ε, επισκόπους και τρεις ε, ιερείς που έχουν απαχθεί στη Συρία και άλλους επίσης που έχουν ε, φωνευθεί. Ο επίσκοπος του Χόμ στις 7 Απριλίου του 2017 δολοφονήθηκε. Μαζί του ήταν άλλος ένας, ο Πατήρ Παορονταλόλιο, που δολοφονήθηκε ε, συγγνώμη, που απήχθη πριν από τρία χρόνια από την Ντάρ στα βόρεια της ε, Συρίας. Αυτή η κατάσταση λοιπόν έφερε την Εκκλησία μας ε, σε θέση να είναι η συνείδηση της κοινωνίας και έμεσα κύριος παράγων, κύριος φορέας, παρά τις εχθρότες και τις καθημερινές δυσκολίε που αντιμετωπίζει αναμφίβολα η δράση της θα γραφτεί μια μέρα στην ιστορία της νέας Συρίας εκείνης που θα κληθεί να αναγεννηθεί και εμφορείται από την Οικουμενική Εκκλησία. Η εμπειρία μου στηρίζεται στην προσωπική μου εμπειρία ως ε, θρησκευτικού άνδρος, ως ιερέως της, ιερέως ε, της Συρίας εμπειρία από το Χόμς και την ευρύτερη περιοχή όπου η Εκκλησία από, μέσω του κλήρου και των διαφόρων ε, έργων που προσφέρει εκλήθη πολλές φορές να παρέμβει για να διαπραγματευτεί ή να διαχειριστεί συγκρούσεις με στόχο να σώσει τη ζωή χριστιανών και μουσουλμάνων χωρίς ούτε μία διάκριση παρά τις ε, λεκτικές απειλές ε, παρά τη λεκτική βία της απειλέ. Δεν δίστασε η Εκκλησία μας να δραματίσει και το ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ των ίδιων των μουσουλμάνων για να μπορέσουν να ανακτήσουν σημεία συνάντησης, για να κλείσουν τα χάσματα που τους διαχωρίσουν. Αυτή η διαπραγματευτική της δουλειά επιστέφθηκε από την απελευθέρωση πολλών ε, αγνοωμένων το Μάιο του 2014 και ήμουν εγώ μέλος της Επιτροπής προέκυψε η ιδέα αυτή από τη δική μας την Εκκλησία και όχι από τα Ηνωμένα Έθνη δεν αποφάσισαν τα Ηνωμένα Έθνη την ε, εκένωση της πόλης της Χόμς και των ε, αντιστεκομένων στις πιέσεις και τις επιθέσεις. Εμείς οι ίδιοι βεβαίως ε, είχαμε αυτή την επιλογή, αλλά ως ήθιστε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, πήραν τη μεγαλύτερη δημοσιότητα. Εμείς όμως ανεβήκαμε στο λεωφορείο, μπήκαμε στο λεωφορείο. Ήμουν ο πρώτος που μπήκε στο λεωφορείο των α, αντιφρονούντων της, ε, μέχρι Χόμς, μέχρι την ιστορική πόλη της Χόμς έτσι ώστε να προσφέρω την εγγύηση πως δεν θα επιτεθεί στο λεωφορείο αυτό ο στρατός, δεν θα πλήξει το λεωφορείο αυτό ο στρατός. Δεν το γνωρίζει αυτό εκείνη η γνώμη. Ε, το 2014 πάλι η Εκκλησία ήταν εκείνη η οποία ανέλαβε τις επαφές, πήρε στα χέρια της επραγματεύσης που επέτρεψαν την ε, απελευθέρωση των ε, αμάχων πρώτα και μετά ε, μαχητών της Χόμς, πρόκειται για την κρίση της παλαιάς πόλης της Χόμς όπως ονομάζεται, που πάλι εξελίχθηκε με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών και όλα αυτά παράλληλα με την στράτευση από την αρχή της Συριακής κρίσης ε, στην προσπάθεια να αποτρέψουμε την εγκαθίδρυση της, ε, του μίσους. Αυτό θέλησαμε να αποτρέψουμε και πώς με κέντρα εκπαίδευσης και κοινωνικής υποστήριξης που προάγουν την ειρήνη μεταξύ των κοινοτήτων θεσπίσαμε ένα κέντρο για τα παιδιά. Με 3.500 παιδιά στη Χόμς και την ευρύτερη περιοχή. Παιδιά προερχόμενα από όλες τις κοινότητες. Παιδιά που είναι οι γονείς τους ακόμη στρατηγοί στο στρατό ή ε, ηγετικά στελέχη των μαχητών της αντίστασης. Ε, αυτός είναι ο μόχθος μας της ε, συνδιαλλαγής και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βλέπουμε ότι διαρκώς προξενούν τη βία για να διχάσουν την κοινωνία της Συρίας αλλά γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά ήδη στη χώρα η εταιρεία του Ιησού και όλοι οι εκπρόσωποι των ε, εγχώριων εκκλησιών από το 2012 κατάφεραν να διασπείρουν κέντρα διαλόγου μέσα από τη δωρεάν παιδεία για τα παιδιά και την κατάρτιση των ενηλίκων απευθυνόμενα σε όλα τα ε, δόγματα και τις ομολογίες και αυτή η εμπειρία συνεχίζεται ακόμη μέχρι σήμερα με βασική αρχή να αγαπάει κανείς τη χώρα του και να εργάζεται για την ειρήνη μεταξύ των κοινοτήτων για να σωθεί η χώρα. Ύστερα από πέντε χρόνια μπορούμε να πούμε ότι έχει φέρει καρπούς αυτή η δουλειά. Είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή, συνεχίζουμε αυτή τη στιγμή να οικοδομούμε μια γενεά της ειρήνης και όχι μόνο παιδιά στρατιώτες ή παιδιά θύματα του πολέμου σε καθαρά ανθρωπιστικό επίπεδο η Εκκλησία συνεργάζεται με τους χριστιανούς και τους μουσουλμάνους χωρίς ουδεμία διάκριση για να φέρουμε την ειρήνη. Έχουμε ομάδες μισές-μισές, χριστιανούς μουσουλμάνους δηλαδή, για να φέρουμε πιο κοντά τα οράματα και να γλυκάνουμε τον πόνο. Τα φιλανθρωπικά χριστιανικά έργα πολλαπλασιάστηκαν, είναι πολλά η δουλειά συνεχίζεται παρά τις δυσκολίες που συγκλονίζουν τη χώρα. Η παρουσία των ακεριοφρόνων δικτύων, των ζυχαντιστικών δικτύων στη Συρία και στο Ιράκ, όπως η Ντάις, Ίσης και Αλνούσρα, δεν ε, βοηθούν μόνο στην καταστροφή της κοινωνίας των ανθρώπων, της θρησκευτική κοινωνίας, η τρομοκρατική δράση της Ίσης δείχνει ότι δεν έχει καμία σχέση με την ε, μουσουλμανική θρησκεία. Θα σας υπενθυμίσω ότι το Ισλάμ συνέβαλε στην ίδρυση του πολιτισμού στη Μέση Ανατολή, ενώ η δράση του ίσης δεν κάνει παρά να διαγράφει κάθε ίχνος πολιτισμού στη χώρα μας. Να σας θυμίσω την καταστροφή των αρχαιολογικών χώρων της Παλμύρας. Μεταξύ άλλων έχει κατεδαφίσει ιερούς ναούς μοναστήρια του 5ου αιώνα, έχει υποχρεώσει χριστιανούς είτε να ε, προσχωρήσουν στο Ισλάμ είτε να πληρώσουν τον κεφαλικό φόρο τους έχει απαγορεύσει την ε, άσκηση των θρησκευτικών τους καθηκόντων πολλοί είναι οι χριστιανοί της Μέσης Ανατολής σήμερα που ε, φοβούνται, αναγκάζονται να φύγουν από τις πατρίδες γιατί φοβούνται νέες εξάρσεις βίας ε, εκθάσεις βίας των οποίων το εύρος διαρκώς διευρύνεται, διαρκώς αυξάνεται. Δυστυχώς πολλοί είναι οι χριστιανοί του εις Βόρειας Συρίας που ήδη έχουν εγκαταλείψει τη χώρα για να πάνε στην Αμερική ή την Ευρώπη. 70% σήμερα των χριστιανών της Βόρειας Συρίας ήδη έχουν φύγει από τη χώρα. Εγώ μιλώ για τη δική μου ε, περιοχή για το δικό μου κλήρο και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το ίμιση των ε, ενωριτών μου βρίσκεται στον Καναδά ή την Ευρώπη και στη Λέσβο που έμεινα τρεις μήνες συνάντησα πάρα πολλούς χριστιανούς που γνωρίζω προσωπικά και που εγκατέλειψαν τη χώρα μας αναζητώντας κάπου στον κόσμο την ειρήνη. Μια κοινωνία λοιπόν με πολυμορφία πολιτιστική και θρησκευτική συνιστά πλούτο. Πολλοί μουσουλμάνοι θέλουν να μείνουν και οι χριστιανοί έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στη χώρα για να οικοδομήσουν την ηθαγένεια που θα αναγνωρίζουν οι πάντες. Δυστυχώς όμως κάποιοι άλλοι θέλουν να, φύγει, να φύγουν οι χριστιανικές κοινότητες. Θα μπορέσουμε να τους επιτρέψουμε να επιστρέψουν. Η δράση σήμερα σημαίνει πρώτα απ' όλα να εξασφαλιστεί η κατάπαυση του πυρός, κοχή. Πέντε χρόνια το λέμε αυτό. Να ενισχυθεί η ειρήνη. Γενέβη ένα, δύο, τρία, δεν έδωσαν κανένα αποτέλεσμα. Ήμουν και εγώ κάπου στις διαπραγματεύσεις Γενέβης, αλλά αντελήφθηνα ότι δεν είναι δυνατόν κανείς να διαπραγματευτεί με ανθρώπους που έχουν γίνει δεκτοί ως διαπραγματευτές, ενώ στην πραγματικότητα είναι ε, ακραίοι, ακεραιόφρονες. Πρέπει να εξασφαλιστεί λοιπόν η συμφιλίωση του Συριακού λαού, πρέπει να εξασφαλιστεί ένα πλαίσιο ανοικοδόμησης. Θα πρέπει να στηριχθούμε στη νέα γενναία, να της δώσουμε από τώρα με την εκπαίδευση, την παιδεία, πάνω απ' όλα την παιδεία, τα μέσα για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Και αυτό πρέπει να αντιληφθείτε, Ευρωπαίοι φίλοι, αγαπητοί Ευρωπαίοι φίλοι. Είναι ότι δεν υπάρχουν μειονότητες στη Συρία. Είναι παγίδα ο όρος μειονότητα. Είναι παγιδευμένος ο όρος μειονότητα. Γιατί αν είναι μειονότητα, αξίζει τον κόπο και να φύγω από τη χώρα, περιμένοντας να με διαγράψει τελείω από το χάρτη η πλειονότητα. Αυτός είναι ο κίνδυνος που ενέχει ο όρος μειονότητα. Μία μόνη μειονότητα υπάρχει στη Συρία. Είναι η Σύρη των διαφόρων ομολογιών και θρησκειών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και, αχ, μιλάω γαλλικά, πώς μου ξεφύγει. Για να ολοκληρώσουμε με τους επισκέπτες μας, ο Πάτερ Εμμανουέλ Γιουκάνα έχει το λόγο. السيدة إلينا فالنسيانو السيدات والسادة أعضاء البرلمان الأوروبي Κυρία Έλενα Βαλεντιάνο, κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, συνάδελφοι, καλησπέρα. Βρίσκομαι εδώ στην Υπεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή πρόσκληση γιατί μιλούμε σήμερα για τις μειονότητες που είναι θύματα του εμφυλίου πολέμου στη ε, Συρία όπως επίσης και από τη βία του Νταέσ ε, στο Ιράκ. Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα το οποίο αφορά τις ε, μειονότητες και όχι μόνο ο ρόλος τους, η ύπαρξή τους απειλούνται ε, μετά από μια ιστορική παρουσία στην Ανατολή και ειδικότερα στη Συρία και στο Ιράκ. Οι χριστιανοί του Ιράκ με την πολιτιστική τους ε, ταυτότητα, τον πολιτισμό τους, πάντοτε ε, είχαν έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Η παρουσία τους, η εκκλησία τους, η πολιτιστική τους παρουσία, είτε είναι Ασσύριοι, είτε είναι Χαλδαίοι, είτε είναι Σύριοι, η η καταγωγή τους είναι αρχαία και σήμερα η ίδια τους η ύπαρξη απειλείται. Πάνω από ένα εκατομμύριο χριστιανοί ε, υπήρχαν στο Ιράκ το 2003, 250.000 έχουν μείνει σήμερα και αυτό που περιμένουμε από τη σημερινή ακρόαση είναι να επιτύχει το γεγονός ότι θα ακουστεί αυτό σε χώρους λήψης πολιτικών αποφάσεων, ε, ώστε να ακουστεί και η δική μας φωνή. Οι Σύριοι είναι εκείνοι ε, που βρίσκονται εκεί με τις ε, υπόλοιπες συνιστώσεις της Συρίας που είναι και εκείνες θύματα της τρομοκρατίας και που αρνούνται την ύπαρξη του άλλου και προσπαθούν ε, να ε, ακυρώσουν την ύπαρξη και ε, την ταυτότητα του. Ζούμε σε αυτό το παγκόσμιο χωριό, τη γη. Υπάρχει τώρα τρομοκρατία που μερικές φορές είναι προέρχεται ε, είναι, προέρχεται από το ISIS, ε, άλλες φορές από, είναι άλλου είδους. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές εκφάνσεις αυτής της τρομοκρατίας. Σήμερα ζούμε την τρομοκρατία του ISIS και αναφέρομαι θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που χαρακτηρίζει τα εγκλήματα του Ισλαμικού κράτους ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας παρόλα αυτά θα ήθελα να επικεντρώσω τη σημερινή μου ομιλία σε δύο βασικούς άξονες. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να περιγράψω αυτήν την τραγωδία, να καταλάβω τους λόγους της και να προσπαθήσω να ε, προτείνω λύσεις. Ε, δεν ε, χρειάζεται, δεν έχει πια νόημα να καταδικάζουμε. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προοπτικές για το μέλλον και για τους χριστιανούς, ώστε να εξακολουθήσει να διαφυλάσσεται η ύπαρξή τους. Θα ήθελα εισαγωγικά να πω ότι δυστυχώς η δίωξη των χριστιανών ε, στην περιοχή δεν ξεκίνησε από τον Τάες και δεν θα ολοκληρωθεί με το τέλος του του Ξεκίνησε με την αρμενική γενοκτονία, τη σφαγή των Χαλδαίων, πάρα πολλές σφαγές που εξακολουθούν να γίνονται και σήμερα. Είναι η φυσική απόρρια, για να το πω έτσι, μιας ε, μη κανονικής ε, κατάστασης. Ε, είναι φυσική απόρρια μιας προσπάθειας ακύρωσης του άλλου ε, όταν ο άλλος είναι διαφορετικός. Ένα ε, περιβάλλον το οποίο υπάρχει εδώ και 1400 ε, χρόνια. τον Νταέσ με τη βαρβαρότητά του, με τη βία του, με τις βίες ματηρές πράξεις, τους, πράξεις του, πρέπει βεβαίως να καταδικαστεί υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να, να καταδικαστούν. Η υποδομή της, ε, των χωρών αυτών, ε, το σχολικό πρόγραμμα, τα καθεστώτα, ε, οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση ακύρωση ε, του άλλου, του διαφορετικού άλλου και δεν υπερβάλλω σε αυτό γιατί το ΝΤΑΕΣ ε, προσπαθεί με άκρο βίαιο τρόπο να ε, επιτύχει αυτό που ήδη υπήρχε στη δομή και στα σχολικά προγράμματα των χωρών της Μέσης Ανατολής. Οι χώρες μας δεν γνωρίζουν την ιδιότητα του πολίτη με την έννοια του να ανήκουμε στο ίδιο κράτος. Πρόκειται για κράτη στα οποία κυριαρχεί ε, το να ανήκει κανείς σε μια συγκεκριμένη θρησκεία και όχι το να ανήκει κανείς σε μια δομή όπως το κράτος. Ε, είναι κάτι το οποίο ισχύει όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο, γιατί μπορεί στη Φαλούτζα κάποιος ή στο ε, Ιράκ να αισθάνεται μια, ότι, ότι μοιράζεται το ίδιο πεπρωμένο με έναν Βόσνιο ή με έναν Ινδονήσιο λόγω του Ισλάμ, ε, λόγω του ότι ανήκει στην ίδια θρησκεία και η οποία ε, αίσθηση είναι πολύ ε, πιο ισχυρή από το γεγονός ότι είναι συμπολίτης με κάποιον Ιρακινό στο Ιράκ. Υπάρχει λοιπόν μια διασυνοριακή αίσθηση του ε, ότι ανήκει κανείς στο Ισλάμ που η κυριαρχή επικρατεί στην έννοια του να ανήκει κανείς στο κράτος του Ιράκ. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο δεν το καταφέραμε. Ε, ε αποτύχαμε να δημιουργήσουμε κράτη που να, δίνουν την αίσθηση μιας εθνικής ταυτότητας και μιας πραγματικής μελλοντική προοπτικής στο πλαίσιο του κράτους αυτού. Και το λέω αυτό και για άλλες χώρες της περιοχής. Ε, συχνά στο Σύνταγμα ο θρησκευτικό νόμο, η Σαρία, κυριαρχεί σε ε, οτιδήποτε στην στη, νομοθεσία ε, την ε, μη θρησκευτική, την κοσμική, οποία δεν μπορεί να κυριαρχεί, δεν μπορεί να επικρατήσει του ε, Ισλαμικού νόμου, γιατί ο Ισλαμικός νόμος κυριαρχεί, επικρατεί, υπερισχύει των υπολείπων νόμων. Υπάρχει έτσι κάπως θεσμοδετείται ε, ε, ε, της, οπότε θεσμοθετείται η, αξία της, της θρησκείας και αυτό έχει αποτέλεσμα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Υπάρχει λοιπόν ένα θεοκρατικό κράτος το οποίο ακυρώνει, εξουδετερώνει τους μη μουσουλμάνους παρά το γεγονός ότι μπορεί να υπήρχαν εκεί πριν από την, από την ύπαρξη του, από την εμφάνιση του Ισλάμ. και Μιλάμε για τις διάφορες ε, κοινότητες του Ιράκ. Θυμόμαστε για παράδειγμα ότι η Σαμπάκ, οι ε, Χαλδαίοι, οι Γεζίντι ε, και άλλες μειονότητες είναι πάρα πολύ παλιές, είναι αρχαίοι λαοί. Υπάρχουν κείμενα που δυστυχώς κυριαρχούν των τωρινών νόμων ε, κείμενα που ε, έχουν μία ε, εντελώς δίσκαμπτη ερμηνεία και είναι κείμενα του ε, παρελθόντος ε, και που δεν επιτρέπουν κατά την ερμηνεία τους το σεβασμό των υπολείπων, ε, όπως επίσης το γεγονός ότι δημιουργούν αυτή την αίσθηση τους Άραβες ότι ήταν πάντοτε αντικείμενο μια συνωμοσία των δυτικών οι Ασσύριοι, οι Χαλδαίοι ε, ήταν πάντοτε ε, θύματα αυτής της ε, συστηματικής πολιτικής στο Ιράκ και στις διάφορες χώρες της περιοχής. Οι χριστιανοί δεν μπορούν πια να περιμένουν. Πρέπει να γίνει κάτι επιγόντως, πρέπει να υπάρξουν προγράμματα υποστήριξης που θα αφαιρέσουν αυτό το αίσθημα απελπισίας και απογοήτευσης και ε, να έχουν μια προοπτική στο μέλλον, να γίνει, σεβαστός ο πολιτιστικό, να γίνει σεβαστή η πολιτιστική τους ταυτότητα, ταυτότητα πριν να είναι πολύ αργά. Πρέπει να διαφυλάξουμε ε, τη σταθερότητα της περιοχής και να προσπαθήσουμε να βρούμε ε, μία λύση προκειμένου να προστατευτούν οι διάφορες κοινότητες. Όσον αφορά συγκεκριμένα το Ιράκ, πρέπει να κάποιες χώρες ε, ε, όπως η Νινεβή και το όρος Σινιάρ να τις απελευθερώσουμε από την παρουσία του Ισλαμικού κράτους και να τους δώσουμε τη δυνατότητα οικονομικής ανάκαμψης. Να δούμε επίση ξανά τις δομές του κράτους ε, σε νομοθετικό και διοικητικό επίπεδο που περιθωριοποιούν τις μειονότητες αυτού, αυτές, να τους δώσουμε ένα ρόλο που να τους αρμόζει και μιλώ κυρίως και για τη δημογραφική παρουσία των Κούρδων στο Ιράκ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η δημογραφία των μειονοτήτων, συγκεκριμένα κυρίως των Γεζίδη και των Χριστιανών, να ε, διασφαλιστεί ε, υπό την αιγίδα του ε, κράτους του Κουρδιστάν, να εξακολουθεί να υπάρχει μια ελευθερία ομολογίας, θρησκείας, ε, μια πολιτιστική ευκαιρία, ε, να μην υπάρχει ένας λόγος που διαδίδει και ενθαρρύνει το μίσος κάθε φορά ε, που οι μειονότητες χάνουν την πίστη στο νόμο, ε, χάνουν την πίστη τους στο μέλλον. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Πρέπει να αναθεωρήσουμε επίσης και τα σχολικά ε, βιβλία, τα οποία δημιουργούν αυτήν την τάση αποξένωσης των μειονοτήτων. Πρέπει να δούμε τον κοινωνικό και εθνικό ιστό στις διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής που αυτή τη στιγμή κατακαιρματίζονται. Υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία δημιουργούν ελπίδα, όπως για παράδειγμα το Κουρδιστάν, γιατί στο Κουρδιστάν 80% των ε, χριστιανών του Ιράκ είναι ευπρόσδεκτη, είναι μια νέα εμπειρία και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε ακόμη εξαγάγει τα απαραίτητα διδάγματα, αλλά είναι κάτι που μπορεί να μας γεμίσει ελπίδα. Και θα ήθελα ε, εν τέλει να ολοκληρώσω λέγοντας ότι κάθε φως είναι καλό, κάθε μικρό κεράκι μπορεί να διαφωτίσει ε, ε, ένα μικρό ε, φως σαν το κεράκι του Κουρδιστάν είναι η λίγη ελπίδα που μας μένει ενδεχομένως. Το ερώτημα λοιπόν που θα ήθελα να ε, θέσω, αυτό που θα ήθελα να ζητήσω από τη διεθνή κοινότητα είναι να υπάρξουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιοχής, όχι μόνο από στρατιωτικής απόψεως, όταν η ε, ε, Πεσμεργά προσπαθούν ε, στα 1500 μέτρα να καταπολεμήσουν το ISIS, ε, πρέπει πραγματικά να ε, προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε την ειρήνη με άλλους τρόπους. Πρέπει να πλησιάσουμε ένα τον άλλον. Οι μειονότητες πρέπει να απελευθερωθούν από αυτή τη φοβία που έχουν έναντι του άλλου έναντι της άλλης ε, ε, μειονότητας και εκεί είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη ευθύνη για όλους όσους έχουν τους σπόρους στα χέρια τους. Πρέπει σε διεθνές επίπεδο να υπάρξει ένα πρόγραμμα διεθνές για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα αποτελεί ένα πλαίσιο αναφοράς. Ε, μας κάνει πολύ εντύπωση όταν βλέπουμε ότι οι χώρες που έχουν κακό ιστορικό παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι αυτές οι οποίες συναλλάσσονται σε εμπορικό επίπεδο με, το, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Συνεχίζει λοιπόν ε, η δίωξη ορισμένων ανθρώπων, η παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητε ποινικέ, οι απαραίτητε οικονομικές κυρώσεις, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία λύση ε, θα έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια θεσμική αντιμετώπιση ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το σεβασμό των μειονοτήτων. Να σα ευχαριστήσω για, τη σημερινή, για την οργάνωση σημερινής ακρόαση και θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι ελπίζουμε ότι ο τρόμος θα σταματήσει και ότι δεν θα φτάσουμε ε, σε, κατάρρευση, σε πλήρη κατάρρευση τη δομή του κράτους. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μπεθέρα θέλει να τη δράσει θα είμαι σύντομη, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που θέλω είναι να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω που ήρθατε. Να σας ευχαριστήσω που για άλλη μια φορά έχετε αυτό το θάρρος να έρθετε και να μας διηγηθείτε πράγματα τόσο δύσκολα, τα οποία χρειάζεται κανείς θάρρος για να τα διηγηθεί. Να μας μιλήσετε για τους μεγάλους, για τα παιδιά που διώκονται, που βιάζονται οι γυναίκες, που σκοτώνονται δικοί τους παιδιά, τα οποία τελικά γίνονται αντικείμενο μίσου. Πράγματι, μερικές φορές και εμείς χάνουμε την εικόνα. Ξεχνάμε. Κι όμως όλοι είμαστε ίδιοι. Τον αναγνωρίζουμε τον άλλον. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε τους ίδιους φόβους, τον ίδιο τρόμο που μας απειλεί. Όλα αυτά πρέπει να πάψουν. Δύο σκέψεις θέλω να σας πω μετά από αυτά που άκουσα. Πράγματι, από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε περιορισμένες δυνατότητες, έχουμε όμως κάποιες δυνατότητες. Πρόσφατα εγκρίναμε ψήφισμα όσον αφορά τη συστηματική σφαγή των θρησκευτικών μειονοτήτων πριν από λίγο καιρό. Το εγκρίναμε. Αναγνωρίσανε πολλές διεθνείς οργανώσεις επίσης και οργανισμοί τη συστηματική γενοκτονία που λαμβάνει η χώρα σε βάρος μειονοτήτων, σε βάρος των Γεζιντή για παράδειγμα. Τώρα από εκεί πέρα, αν υπάρχει κάτι στην πράξη που μπορούμε να κάνουμε, αυτό είναι ότι έχουμε τη συμφωνία για τη γενοκτονία και πώς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα επιληφθεί. Υπάρχουν στοιχεία. Αυτά πρέπει να φτάσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο νομικά επεξεργασμένα με τον καλύτερο δυνικό τρόπο, ώστε να προχωρήσει αυτή η υπόθεση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και εμείς από και πέρα από τις χώρες μας, να πιέσουμε τις κυβερνήσεις μας, μια που και εμείς συμμετέχουμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύω ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν μη τι άλλο συμφωνούμε γι' αυτό, για αυτά που ακούσαμε σήμερα. Οπότε έχετε το σεβασμό μου. Σας λέω ότι είμαι διατεθειμένη να δουλέψω προς αυτή την κατεύθυνση για να βοηθήσω στην πράξη όσο γίνεται την υπόθεση σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ που ήρθατε να μας μιλήσετε. Έχω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις, κυρία Τάρ, πρώτα εσείς. Αν κατάλαβα καλά τα λόγια σας, Είπατε ότι έχουν ε, προβλήματα σε σχέση ε, και με τη διαμονή τους στη Γερμανία οι Γεζιδίτες. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό. Και δεύτερον, για τον το Ιουκάνα. Όπως ρώτησε και η προηγούμενη συνάδελφος, νομικά τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Πρακτικά, παραδείγματι, προσφερόντας βοήθεια, ή κάτι άλλο. Ξέρετε ότι ως Κοινοβούλιο έχουμε πολύ πολύ περιορισμένες δυνατότητες. Πάντως υπάρχουν κάποιες δυνατότητες που θα μπορούσαμε ίσως ε, από εσά να εμπνευστούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ένα λεπτό καθένας για να απαντήσει. Αλλά προηγουμένω να ξέρω κατά πόσο ο εκπρόσωπος από την υπηρεσία για το Ιράκ θέλει το λόγο. Παρακαλώ η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στο τμήμα που είναι αρμόδιο για το Ιράκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Γκάι Χάρισον ονομάζομαι. Και όντω είμαι στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης υπεύθυνο για το Ιράκ. Αυτά τα οποία ακούσαμε είναι πράγματα με τα οποία είμαστε δυστυχώς εξοικειωμένοι. Τις τραγωδίες τις έχουμε ακούσει και στο Ιράκ και στη Συρία. Η κατάσταση των μειονοτήτων στο Ιράκ αποτελεί και το βαρόμετρο για την κατάσταση σε όλες τις γείτονε χώρες. Για την ανθρωπιστική βοήθεια, για τις διώξεις, για την κατάσταση όσον αφορά τη δημοκρατία στις χώρες αυτές. Θέλω να υπογραμμίσω ότι για μας, όχι μόνο δηλαδή για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την αντιπροσωπεία της στο Ιράκ, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΟ, την ΤΕΦΚΟ, παρακολουθούμε αυτές τις υποθέσεις από κοντά όσο μπορούμε και σε επίπεδο χωρών μελών επίσης. 23 Μαΐου θα είδατε τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ε, πάντα επαναλαμβάνουμε στην πρώτη παράγραφο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται για την ε, ελευθερία θρησκείας και στο Ιράκ και στη Συρία και στην περιοχή γενικότερα. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε. Το πρώτο που πρέπει εδώ να υπογραμμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη συλλογικά είναι κύριοι δωρητέ στη Συρία και το Ιράκ. Όμω, δεν σημαίνει ότι τα πράγματα είναι καλά. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα ανθρωπιστικά σχέδια του ΟΗΕ για την διεθνή κοινότητα χρηματοδοτούνται μόνο σε ένα 30%. Έτσι καλύπτονται οι βασικές ανάγκες, αλλά τα, όλα τα υπόλοιπα δεν καλύπτονται δυστυχώς. Δουλεύουμε λοιπόν μέσω της αναπτυξιακής βοήθειας και άλλων πόρων που συλλέγονται για να βοηθήσουμε τις μειονότητες, κυρίως αυτές που αποτελούν πιο πολύ στόχο με προγράμματα ώστε να στηρίξουμε και να προστατεύσουμε τα δικαιώματά τους. Υπάρχει συμφωνία συνεργασίας στο Ιράκ για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμφωνία που έχουμε δηλαδή με την κυβέρνηση του Ιράκ. Δύο συναντήσεις είχαμε μαζί τους μέχρι τώρα. Αυτό που πρέπει να υπογραμμίσω, και βέβαια δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε δεδομένο σε μια περιοχή όπου οι κυβερνήσεις συχνά δεν είναι διατεθειμένες, δεν είναι πρόθυμες να μιλούν για ανθρώπινα δικαιώματα, είχαμε επικοδομητική συζήτηση με την κυβέρνηση του Ιράκ. Θέλουμε όμως βέβαια να δούμε περισσότερες δεσμεύσεις και ακόμα περισσότερες δράσεις ε, στους διαλόγους αυτούς. Στηρίζουμε το Ιράκ και τις μειονότητες εκεί, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις περιοχές τους με το σχέδιο σταθεροποίησης από πλάση του ΟΗΕ και θα σας δώσω λεπτομέρειες αν επιθυμείτε αργότερα. Τώρα για τους ε, Γεζιντή. Βεβαίως και θέλουμε να υποστηρίξουμε κάποια δράση επρόκειτο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, δεν υπάρχει αμφιβολία. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι τα εγκλήματα αυτά έλαβαν χώρα. Η ευρωπαϊκή εμπειρία, για παράδειγμα μετά από την Βοσνία, στην τέως Ιουγκοσλαβία, ξέρουμε ότι χρειάζεται χρόνος ε, κυβερνήσεις να συνεργαστούν για να φτάσει ο φάκελος στο ποινικό δικαστήριο. Πρώτα περνάει από τα εθνικά δικαστήρια και μετά πάει στο διεθνές. ζητήσατε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συγκέντρωση στοιχείων. Το ξέρω, το έχουμε πάρει το αίτημα, το εξετάζουμε. Μέχρι τα τέλη της χρονιάς θα ξέρουμε περισσότερα. Γίνεται δουλειά τώρα που μιλάμε. Ξέρουμε ποιο είναι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που στηρίζει τα θύματα των εγκλημάτων αυτών. τονίζουμε ότι έτσι καλώς η επανόρθωση αφορά την νομική πτυχή και όχι τις πραγματικές ανάγκες των θυμάτων. Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε εμείς να προωθήσουμε. Αλλά εξαρτώμεθα και από την Ιρακινή κυβέρνηση. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις που έχουν φτάσει στην Ιρακινή κυβέρνηση και περιμένουμε την απάντηση τώρα του Ιράκ. δεν θέλω να μακρηγορήσω. Αν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα ζητήματα, ευχαρίστω να σας απαντήσω. Στήριξη δίνουμε. Εντάξει, ξέρω ότι αυτό δεν είναι παρηγοριά για αυτούς που υποφέρουν από τρομερά εγκλήματα σαν και αυτά της ΔΑΕΣ. Η ΔΑΕΣ είναι ένα στρώμα του προβλήματος. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά στρώματα, πολλές στιβάδες πρέπει να συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στο Ιράκ και τα επόμενα χρόνια, για πολύ. Όχι μόνο μέχρι το 2016, τώρα κοιτάμε να δούμε τι θα κάνουμε μετά το 2016, τι πολιτική θα ακολουθήσουμε και βέβαια χρειαζόμαστε και τους ανάλογους πόρους για να την υλοποιήσουμε. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε πολύ για τις επεξηγήσεις. Ερωτήσεις προς τον ε, εκπρόσωπο υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είπα ακριβώ αυτό. Ίσως δεν με καταλάβατε καλά. Από τη διεθνή κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ζητάμε τίποτα άλλο από τα δικαιώματά μας. Αν δεν ήμασταν σε τόσο τραγική κατάσταση, δεν θα όργανα όλο τον κόσμο στώντας ε, βοήθεια. Είμαστε μια πολύ μικρή μειονότητα, έχουμε πέσει θύματα γενοκτονίας διαχρονικά. Χιλιάδες κορίτσια στο Ιράκ και τη Συρία πέφτουν θύματα βιασμών από το ΙΣΙΤ. Και δεν έχουμε λάβει την παραμικρή βοήθεια ούτε στο Ιράκ, ούτε στο καν στο Κουρδιστάν. Η ίδια μας η χώρα δεν μας προστάτευσε στο Μπίλεφελτ της Γερμανίας τι συνέβη. Αφγανοί και Σύριοι επτέθησαν κατά Ιαζιδιτών με χμηρά αντικείμενα μαχαίρια φωνάζοντας είσαστε άπιστοι. Από αυτό προσπαθούμε να γλιτώσουμε. Δεν είμαστε εμείς σαν αυτούς που φύγαν από τις χώρες τους εξάγοντας και την τρομοκρατία μαζί τους. Ο κύριε Σεβασμιότητος Γιουκάνα, Ναι, ευχαριστώ κύριε Μπούχνερ. Είμαι διευθυντής φιλανθρωπικής οργάνωσης στο Ιράκ και γνωρίζω καλά τις ανάγκες τι χρειάζεται για να σωθεί μια ζωή, τι, τι χρειάζεται ως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ως παιδεία, ως πρόγραμμα αποκατάστασης, ανοικοδόμησης. Τα γνωρίζω όλα αυτά. Αγαπητοί φίλοι όμως, αυτό που χρειαζόμαστε είναι κάτι που ξεπερνά την ηλική υποστήριξη. Οι Ασσύριοι, οι Χριστιανοί, οι Γεζιδίτες είναι τα θύματα μίας καταστροφής που έχει προκαλέσει ο ίδιος ο άνθρωπος. Αυτό που ζητούν είναι να ανακτήσουν την αξιοπρέπειά τους, να εξασφαλίσουν την ύπαρξή τους την ίδια, τη διαιώνιση των κοινοτήτων τους στη χώρα τους. Και όπως είπα και στην ομιλία μου, πρέπει να επανεξεταστούν τα σχολικά εγχειρίδια, οι οδηγοί σπουδών, νομοθεσία. Εγώ απευθύνω εκλειστό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς να γνωρίζω τις ιδιαιτερότητες των αρμοδιοτήτων του ενός ή του άλλου. Σας καλώ όμως να επικοινωνήσετε με τις κυβερνήσεις σας και να ζητήσετε να δοθεί μια απάντηση στις προσδοκίες μας, όχι μόνο ως υλική υποστήριξη, αλλά πέραν αυτής η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Κύριε Άντριος, για να έχουν όλη την ευκαιρία να απαντήσουν. Συνεχίζοντας ε, τις ερωτήσεις που άκουσα και να πω και κάποια πράγματα που δεν είπα προηγουμένως, υπάρχει, υπάρχουν τα βραχυπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν. Βράχυπρόθεσμα χρειάζεται περισσότερη στήριξη για να προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι στο Ιράκ και χρειάζονται περισσότερε προσπάθειε ώστε να υπάρξει μια κατάσταση ασφαλεία σε απελευθερωμένε περιοχέ που δίνουν τη δυνατότητα στι μειονότητε να νιώσουν ότι μπορούν να γυρίσουν πίσω στα σπίτια του. Για την ώρα οι άνθρωποι είναι πολύ καχύποπτοι ε, προς τους ε, ε, Κούρδους αντάρτες τους Πεσμερικά, προς τον στρατό, ομάδες οι οποίες στο παρελθόν έδρασαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παίρνουν ολόκληρες περιοχές από τις μειονότητες αυτές και προσπαθούσαν να περάσουν τη δική τους ε, ε, θεώρηση του τι ακριβώς σημαίνει Ιράκ για εκείνους. Θα ήθελα να υπάρξει λοιπόν περισσότερη υποστήριξη ε, της κοινωνίας των πολιτών, ώστε οι μειονότητες να έχουν μία φωνή που θα εισακούεται και δεν θα χρειάζεται να έρθουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους. Πρέπει να σταματήσουμε τα μέτρα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση στο Ιράκ, δηλαδή να προσπαθούν να φημώσουν μέσα ενημέρωση που προσπαθούν να υποστηρίξουν τις ε, ομάδες αυτέ. Ε, όπως επίσης και το κυβερνητικό ε, στρατό, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που τώρα είναι υπό τον έλεγχο ορισμένων συγκεκριμένων ομάδων και της κυβέρνησης του Ιράκ ε, να ε, μπορέσουν ε, να δώσουν τη δυνατότητα στις ομάδες των μειονοτήτων να ακούγονται καλύτερα, να εισακούονται καλύτερα και να έχουν τη θέση τους στην κοινωνία του Ιράκ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω το εξής. Σήμερα αναφέρθηκα σε όλες τις ευάλωστες ομάδες στο Ιράκ. Δεν μπορούμε να επικεντρωνόμαστε σε μία συγκεκριμένη ομάδα και να γνωρούμε τις υπόλοιπες ε, Ζητά ο ε, συνάδελφος ε, την ενίσχυση των ε, χριστιανών. Όμως το 1 τέταρτο της, του εδάφους του Ιράκ είναι στα χέρια του Άιζες, Αυτό είναι το πρόβλημα. Πάνω από 4 εκατομμύρια άτομα είναι εκτοπισθέντες. Δεν είναι μόνο γεζίδις και χριστιανοί. Ε, αυτό που γίνεται τώρα με αυτές τις ομάδες είχε αρχίσει και με τους, ε, είχε γίνει και στους Ουρκομάνους. Μην ξεχνάμε τι είχε γίνει ε, με την πόλη φόρο όταν χρειάστηκε να φύγουν τόσες, τόσες χιλιάδες Τουρκομάνοι. α, όλες οι, οι, οι, ομάδες, όλες οι μειονοτικές ομάδες που υπέστησαν αυτήν την κατάσταση από το ISIS πρέπει να υποστηριχθούν ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια τεράστια τρομοκρατική απειλή αυτή τη στιγμή στο Ιράκ, ανεξαρτήτως εθνότητας, ανεξαρτήτως ε, θρησκείας. Ε, υπάρχουν τεράστιες συνέπειες για όλους και πρέπει να, να υποστηριχθούν όλες αυτές οι ομάδες με, με ε, όμοιο τρόπο, ανεξαρτήτως εθνότητας και θρησκείας από τη διεθνή κοινότητα και συμφωνώ με τον συνάδελφο, πρέπει να ενισχύσουμε την κοινωνία των πολιτών στο Ιράκ, ώστε οι άνθρωποι, οι, οι, οι, οι πολίτες, ε, οι μειονότητες να ε, μπορούν να υπερασπιστούν τον ε, εαυτό τους χωρίς να χρειάζεται να έρχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να το κάνουν. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να σας ευχαριστήσω όλες τις κυβερνήσεις σας ε, που κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, όμως στο Ιράκ χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Εσείς τώρα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία που έχει η ανθρωπιστική βοήθεια για τη Εκκλησία στη Συρία. Γιατί όπως σας εξήγησα, η εκκλησία παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο για να συνεχιστεί το εκπαιδευτικό έργο, αλλά και να αντιμετωπιστούν οι επιτόπου προκλήσεις. Δεν πρόκειται μόνο για συνεργασία με τον Ερθρό Σταυρό ή άλλους, κάνουν και αυτή τη δουλειά τους βέβαια, για την διατροφή, για την υγεία, αλλά μην ξεχνάμε και την εκπαίδευση γιατί μόνο τότε μπορούμε να έχουμε μια καλή νέα γενιά. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να πούμε ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε με τους ανθρώπους που κάνουν τις διαπραγματεύσεις στη Συρία. Το κυβερνήτη της Χόμς ή εμένα τον ίδιο συνεργάστηκα μαζί του. Η αποστολή, το ίδιο επίσης συνεργάζονται μαζί του και έχει το σεβασμό όλων. Τρίτον, σύντομα, Μέχρι σήμερα δεν καταλαβαίνει κανείς ο Σύριος ή Ρακινός πώς ένας στρατός τόσο ισχυρός όπως αυτός του Σαντάμ Χουσέιν μέσα σε δυο μέρες σητήθηκε. Και δεν καταφέρνουμε να ξεγράψουμε την ΤΑΕΣ εδώ και τόσο καιρό. Ρωτάνε ο κόσμος τι κάνει το ΝΑΤΟ σήμερα. τελικά ε, γίνονται σπατάλες. Τι γίνεται, οι... τα βλήματα πέφτουν δεξιά-αριστερά χωρίς να στοχεύεται πραγματικά την ΤΑΣ. Ποιος τους χρηματοδοτεί με τέτοια τεχνολογία που έχετε, σκέφτεται ο κόσμος, με τις νέες τεχνολογίες. Πώς δεν τα καταφέρετε με τόσες υπηρεσίες πληροφοριών που έχουν τις νέες τεχνολογίες στα χέρια τους. Συνεπώς πρέπει να δράσουμε, δεν μπορεί να αφήνουμε την ΤΑΕΣ που έχει ένα κράτος το οποίο είναι εντελώ φτιαχτό. Εμείς δεν είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια τρομοκρατική οργάνωση. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Να ξέρετε ότι εμείς δεν τα βάζουμε με κανέναν και εμείς δεν σπέρνουμε βλήματα δεξιά-αριστερά. Αυτά. Λοιπόν, πρώτον, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ και για το καθημερινό σας έργο, γιατί εσείς έρχεστε εδώ, σας δίνουμε εδώ 12 λεπτά για να μας εξηγήσετε μερικές φορές την ίδια σας τη ζωή ολόκληρη. Το ξέρετε ότι είσαστε απαραίτητοι σε αυτή τη διαδικασία, ελπίζουμε, εθνική συμφιλίωσης στις χώρες εκείνες για τις οποίες μιλήσαμε σήμερα. Αυτά που μας είπε ο Σεβασμιότατος για το Κουρδιστάν είναι πράγματα, ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες περιοχές για να δείχνουμε κατανόηση και να σεβόμαστε τον άλλον. Και φυσικά η εκπαίδευση έχει πρωτεύοντα ρόλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις πρωτοβουλίες σας. Εντάξει, δεν είναι αυτό που μας φτάνει, αλλά όπως είπε πριν και η κυρία Μπεθέρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμευόμαστε υπέρ του δικού σας αγώνα. Και το πρωταγωνιστικό ρόλο τον έχετε εσείς. Εσείς θα οικοδομήσετε την ειρήνη. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που ήρθατε εδώ. Σας ευχαριστούμε όλους. Θα συνεδριάσουμε και πάλι 15 Ιουνίου, πρωί και απόγευμα.